Okay, colleagues, we wait a little bit because we know it's Monday. Συνάδελφοι, περιμέναμε λίγο γιατί ξέρουμε ότι είναι Δευτέρα, κάποιοι συνάδελφοι ταξιδεύουν, αλλά θα ξεκινήσουμε. Ε, σιγά σιγά. ξεκινάμε γιατί έχουμε και πολλά στην μέσα διάταξη. Ε, σημείο 1. Υπάρχει μια τροποποίηση της μέσης διάταξης. Που είναι η εξής. Το σημείο 23 και 24 ε, θα τα εξετάσουμε πριν από το 22. και μετά θα περάσουμε στη κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, θα κλείσουμε μάλλον τα ζητήματα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή και τα διάφορα πριν περάσουμε στην άλλη συνεδρίαση, αύριο το απόγευμα. Και υπάρχει και μια άλλη τροποποίηση, δεν έχω εδώ βέβαια τους αριθμούς. Το σημείο 8 της Heidi Hautala. Το ανταλλάσσουμε με το σημείο 21, την κατάσταση στο Ιράκ, του κυρίου Βάιρενεν. Γιατί η κυρία Χάουταλα δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα εξετάσουμε λοιπόν το δικό της θέμα αύριο το απόγευμα. Ανταλλάσσουμε λοιπόν το 8 με το 21. Συμφωνείτε με τη μεσαία διάταξη. Ωραία, ευχαριστώ. Ανακοινώσει της Προέδρου με την ιδιότητα του Συμπροέδρου της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσως Εκπροσώπησης ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Λουί Μισελ ξεκίνησε ένα ε, έργο για νέα στελέχη για να εξοικειωθούν με τα λεγόμενα μυστήρια των, ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, σκηνής. Εντάξει, ας μην τα κάνουμε. Ας μην ανακοινώσουμε τώρα τους καλεσμένους μας που έρχονται από την ε, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Θα το κάνουμε στην πορεία. Υπερθυμίζω ότι αύριο θα γίνει μια ειδική συνεδρίαση με την Επιτροπή ΙΝΤΑ στις 11.30 το πρωί. Και την Τετάρτη το πρωί έχουμε και μια ειδική συνεδρίαση με την Concord, το συνασπισμό και στην Ομοσπονδία μάλλον των ε, ΜΚΟ. Θα εξετάσουμε το επερχόμενο πολιτές νομικό πλαίσιο, το μέλλον της εταιρικής σχέσης ε, με το Κοτονού ε, και τα εχέγγυα της δικλήτης ασφαλείας κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ούτω καθεξής. Αυτό θα γίνει αύριο στις 10, από τις 10 έως τις 12.30. Ελπίζω τα μέλη μας να είναι εκεί. Έχω μερικές θετικές ειδήσει για το προσωπικό μας. Ο Γέσπερ Χάγκλουντ έχει επιστρέψει. Ε, πέρσι έφυγε, πήγε στο επιτελείο του Προέδρου και τώρα επέστρεψε στην Επιτροπή μας. Τον ευχαριστούμε που επανήλθε. Καθώς ε, υποδεχόμαστε και την Τζουλιέτα Μπιντήλη, Βοηθό πλέον στην ομάδα μα, στην Επιτροπή μα, καλώ ήρθε, Και ο Νίκολα Στεφανούτα. Είναι εδώ. Όχι. Ήταν στην ΤΕΒΕ για μερικού μήνε, Τώρα ε, έφυγε. Ε, θα περάσει μερικού μήνε στην Επιτροπή Ντρουά πριν ε, μεταβεί στην Ουάσιγκτον. Αυτέ είναι οι αλλαγέ λοιπόν επί του προσωπικού. Περνούν στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 19 και 20 Φεβρουαρίου τα έχετε στου φακέλου, Αν υπάρχουν σχόλια, παρακαλώ να μα ενημερώσετε μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση. Ιδάλω θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Τα πρακτικά της 27 η Φεβρουαρίου θα τα εγκρίνουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Τέσσερα. Ε, αποφάσεις και συστάσει των συντονιστών. Έχετε ε, τα σχετικά έγγραφα της 20ης Μαρτίου στους φακέλους και πάλι αν έχετε σχόλια παρακαλώ στη γραμματεία. Ιδάλλως ε, θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Σημείο 5. Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο πρώτο ουσιαστικό σημείο της μεσης το σημείο 6. Μια ανταλλαγή απόψεων με τον Μαρκ Λόκοκ, Γενικό Υπογραμματέα του ΟΗΕ ε, για ανθρωπιστικά ζητήματα και ε, για την παροχή έκτακτης ε, βοήθειας και είναι και επικεφαλής του Γραφείου Συμπενισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων της ΟΤΣΑ. Χαίρομαστε διατέλους που έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Ξέρουμε ότι είστε εδώ για μια πολύ σημαντική συνδιάσκεψη για τη Συρία που θα γίνει τις επόμενες δύο ημέρε στις Βρυξέλλες. Για να σας δώσω λίγο μια εικόνα για τον Λόκοκ. Ε, ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου του 2017, ε, μετά τον Στίβεν Ομπράιεν που είχαμε γνωρίσει την προηγούμενη φορά. Προηγουμένω, ο κ. Λόκοκ ήταν μόνιμος ε, γραμματέας ε, του Ευρωπαϊκού Υπουργείου Διεθνούς Ανάπτυξη, DFIT, και εδώ και πάνω από 30 χρόνια εργάζεται σε αυτόν τον τομέα της διαχείρισης και συντονισμού ε, ανταπόκρισης ε, και παροχής έκτακτης βοήθειας σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Θα σας δώσω απευθείας το λόγο. Να πω μόνο ότι έχουμε λίγα μέλη εδώ. Είναι ο κύριος Νόιζερ, Βέντε, εκπροσωπούν τις δύο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, το ΕΛΚ και τους Συλλογιστές Δημοκράτες και σίγουρα θα έρθουν και άλλοι στην πορεία. Παρακαλώ. Well, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά να εδώ σήμερα. Ε, είμαι με την ιδιότητα που έχω στον ΟΗΕ, είμαι αρμόδιος για ζητήματα παροχής ε, βοήθειας, ε, όχι μόνο στον ΟΗΕ, αλλά γενικότερα στο σύστημα ε, παροχής ανθρωπιστική βοήθειας και ΜΚΟ και το καθεξής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος υπέρμαχος της ανθρωπιστικής ε, δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από εσάς δηλαδή συλλογικά. Τα όσα κάνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα κράτη-μέλη ε, σας καθιστούν ε, τον μεγαλύτερο χρηματοδότη ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον κόσμο. Και σας ευχαριστώ και εσάς και τους ψηφοφόρους σας για αυτή τη στήριξη. Να πω δύο λόγια, αν με επιτρέπετε, ε, εν είδη αξιολόγησης του ανθρωπιστικού συστήματος ε, παγκοσμίω αυτή τη στιγμή και θέλω να σταθώ και σε τις μεγάλες προκλήσεις και κρίσει που αντιμετωπίζουμε και μετά να αναφέρω και ορισμένες μελλοντικέ προοπτικές ε, και τον κεντρικό ρόλο που θεωρώ ότι θα διαδραματίσει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας για την υλοποίηση αυτών των νέων ευκαιριών. Το ανθρωπιστικό σύστημα είναι πιο αποτελεσματικό από ποτέ. Κάθε χρόνο ε, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, φτάνουν σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων και σώζουν εκατομμύρια ζωές. Το έχω δει και με τα μάτια μου στις χώρες που έχω επισκεφθεί. Ε, το τελευταίο χρόνο έχω επισκεφθεί τη Συρία, τη Σομαλία Έχω δει τους ε, Ροχίνια που φύγαν από την ε, ε, Μιανμάρ, Σομαλία, Αιθιοπία, μιλήσαμε για τη, δημοκρατία, τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό που πήγα προσφάτως, Σουδάν και Νότιο Σουδάν. Όπου πηγαίνω βλέπω εκατοντάδες φορείς με εκατοντάδες και χιλιάδες ε, υπαλλήλους προσωπικό που καλύπτουν τις ανάγκες του κόσμου εκεί και πέρα από τι προσπάθειε που διευκολύνονται, μάλλον χωρί αυτή την βοήθεια, χωρί αυτή την παρουσία την οποία διευκολύνεται και εσεί, θα χάνονταν εκατομμύρια ζωέ. Πέρσι λοιπόν καταφέραμε να αποφύγουμε λοιμούς ε, στο Νότιο Σουδάν, στην Ιεμένη και σε άλλες χώρες. Ε, βοηθήσαμε τους Ροχίνγκια Έχουμε και τους εκτοπισμένους ε, σε όλο τον κόσμο, από την Κολομβία μέχρι την Ουκρανία. Επίσης, ε, είμαστε καλύτεροι να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες. Ε, συντονισμός και συνεργασία μεταξύ της πρωτοβάθμιας παροχής βοήθειας και των υψηλότερων, πιο υψηλόβαθμων φορέων. Υπάρχει βελτίωση σχέση με το παρελθόν. Οπότε το κάθε ευρώ δαπανάται και πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικά προκειμένου να σώσουμε ζωές. Όλα αυτά λοιπόν ισχύουν. Από την άλλη όμως ε, φαίνεται ότι οι ανάγκες ε, αυξάνονται κάθε χρόνο και ότι ζητούμε περισσότερα χρήματα κάθε χρόνο. Έτσι λένε ορισμένοι. Και τίθεται το ερώτημα Πώς γίνεται αυτό. Και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα γιατί πρόκειται για παράδοξο. Αφενό τα τελευταία 40-50 χρόνια 100 χώρες ανά τον κόσμο έχουν ε, ε, προοδεύσει σημαντικά και οικονομικά και κοινωνικά. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, ε, έχει πέσει η θνησιμότητα παιδιών. Από την άλλη όμως 30-40 χώρες δεν έχουν δει αυτή την ε, πρόοδο, κυρίω στην Αφρική και την ε, Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν έχουν αυξηθεί οι ανθρωπιστικές ανάγκες σε ορισμένε αυτές τι χώρε. Πέρσι και φέτος εμείς ε, στον ΟΗΕ και σε κλίση που έχουμε απευθύνει έχουμε ζητήσει ποσά ρεκόρ για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που εξηγούν γιατί παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια, έχουμε λοιπόν τρεις βασικές αιτίες που εμείς ζητούμε περισσότερα κονδύλια τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, έχει αυξηθεί κατά ένα δις ο ανθρώπινος πληθυσμός σε σχέση με το 2005. Και περισσότεροι από αυτούς, τους ανθρώπους, ε, ζουν σε χώρες ε, υψηλών ανθρωπιστικών αναγκών. Δεύτερον, έχουμε ένα κύμα ε, τρομερών συγκρούσεων, ιδίως μετά το 2010, ιδίως στη Συρία, που όπως είπατε και εσείς ε, είναι ένας τους λόγους που με εδώ στις Βρυξέλλες, αν και θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς, γιατί θέλω να σας δω. Στην Ιεμένη, Ιράκ, στο σύνολο της Αφρικανικής Υπήρου, Αυτές οι συγκρούσεις κάποιες φορές οδηγούν σε ε, τρομοκρατία και έχουν ε, οδηγήσει τεράστιες ε, ανάγκες. Γενικά, επίσης, έχουν αυξηθεί και τα πρότυπα σε τη φορά την ανταπόκριση και την παροχή βοήθειας. Εγώ, α πούμε, τη δεκαετία του 80 ασχολούμουν ιδίω με την Αιθιοπία. Τότε θέλαμε τροφή, νερό και καταφύγιο. Τώρα όμως έχουμε ε, υψηλότερες απαιτήσει, πρόσβαση στο σχολείο, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, βιωτικό επίπεδο, εισόδημα. Και αυτό είναι θετικό που έχουμε γίνει πιο φιλόδοξοι και πιο αποτελεσματικοί, γιατί θέλουμε ουσιαστικά να ε, βελτιώσουμε τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Έχουμε μία σειρά τρόπους για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Πρώτα πρέπει να δούμε τον τρόπο χρηματοδότησης των ανθρωπιστικών κρίσεων. Αυτή τη στιγμή, το λέω είναι ήδη καρικατούρας, αλλά όχι και τόσο τελικά, βλέπουμε ότι ο κόσμος παρακολουθεί καθώς γύρεται ένα νέο πρόβλημα ε, δημιουργείται μια αίσθηση της κοινή γνώμης, οι πολιτικοί θεωρούν ότι πρέπει να ανταποκριθούν, κινητοποιούνται κονδύλια και οι φορείς ε, δραστηριοποιούνται. Αυτό συνήθως παίρνει πολύ χρόνο. Για τις περισσότερες από τις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, είτε πρόκειται για σεισμούς, πλημμύρες, ξηρασίες και άλλες φυσικές καταστροφές, γνωρίζουμε ότι θα προκύψουν. Μπορεί να μην ξέρουμε πότε ακριβώς θα συμβεί ο επόμενος σεισμός ή πότε θα έρθει η επόμενη ξηρασία. Γνωρίζουμε όμως ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον πλανήτη μας και μπορούμε να αναπτύξουμε συστήματα ανταπόκρισης που θα είναι καλύτερα σχεδιασμένα για να ε, προκαταλαμβάνουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε καλύτερη χρήση ασφαλιστικών μηχανισμών. Τις πρώτες εβδομάδες ε, που ανέλαβε τα καθήκοντά μου, ε, συντόνιζα την ανταπόκριση για τους ε, κυκλώνε και τους τυφώνε στην Καραϊβική. Ευτυχώ αυτή η διαδικασία πήγε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Μέσα σε μερικές μέρες και εβδομάδες καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τους πόρους. Αντίστοιχα, μπορούμε να κάνουμε καλύτερη χρήση των δεδομένων έγκαιρη προειδοποίηση και αντίστοιχων δικτών για να κινητοποιούμε πόρου πιο γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε ξηρασίες. Ξέρουμε ότι σε ορισμένες χώρες θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτε και συστηματικά θα είναι ευάλωτε στι ξηρασίες, ιδίω και εξαιτία τη ε, κλιματική αλλαγή. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ε, με βάση τα στοιχεία που εξετάζουμε εμείς, τους δείκτες που εξετάζουμε, να περιμένουμε μέχρι το σημείο που ε, η περίμετρος ε, του μπράτσου ενός παιδιού θα είναι τα δεκατοστά πριν αναλάβουμε δράση. Πολλά περισσότερα μπορούμε να κάνουμε και για να συντονίσουμε καλύτερα την ανθρωπιστική βοήθεια. και υιοθετήσετε και σε ένα ψήφισμα πριν από μερικέ εβδομάδε, όπου εξετάζετε την ανάπτυξη ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια και σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Εξέτασα το κείμενο, το οποίο είναι καλό. Και πολλά από αυτά που αναφέρετε μας βρίσκουν σύμφωνους. Θεωρούμε και εμεί ότι πρέπει να υιοθετήσουμε αυτά τα στοιχεία, ιδίως ε, για την ανθρωπιστική ανάπτυξη. Στη Σομαλία, για παράδειγμα, όπου τα τελευταία 25 χρόνια έχω περάσει πολύ καιρό. Πέρυσι, για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο λοιμού, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα ε, μεταβίβασης ε, μετρητών και έτσι 3 εκατομμύρια ε, άνθρωποι έλαβαν κάποια χρήματα για να αποφύγουν την κρίση. Ξέρουμε ότι θα ανακύψουν φαινόμενα ξηρασία στη Σομαλία. Επομένως, Έχουμε δημιουργήσει αυτή τη πλατφόρμα, πρέπει λοιπόν να τη διατηρήσουμε, ώστε την επόμενη φορά που θα έχουμε μια ξηρασία οι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε ήδη έχουν καταχωριστεί στο σύστημα και θα μπορούν να λάβουν πιο σύντομα ένα μικρό έστω ποσό σε σχέση με προηγούμενες τις περιπτώσει. Αυτά τα συστήματα κοινωνική προστασία έχουν ε, δημιουργηθεί ήδη σε μία σειρά χώρε και μπορούν να συσταθούν και σε άλλε χώρε όπω η Σομαλία και η Εμένη. Να σας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα. Πολύ συχνά οι ανθρωπιστικοί φορείς ε, δαπανούν χρήματα απλώ για να μεταφέρουν νερό από τη μια περιοχή στην άλλη. Καλό θα ήταν να συνεργαστούν ε, και να επενδύσουν στην καλύτερη διαχείριση υδάτων για να μην φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα καλύτερης, ε, καλύτερης συνεργασίας μεταξύ του ανθρωπιστικού κλάδου και του αναπτυξιακού κλάδου. Ε, έχω συνεργαστεί με πολλές οργανώσεις που αντιμετωπίζουν και το ανθρωπιστικό και το αναπτυξιακό σκέλος. Ε, είμαι ιδιαίτερο υπέρμαχο όλων αυτών και ο κύριος Γκουτιέρες έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε όλα αυτά στην προσέγγιση του για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ μπορούμε να γίνουμε και πιο αποτελεσματικοί και ως προς το κόστος αν θέλετε και χαίρομαι που το εντοπίσατε στο έγγραφό σας γιατί ξέρουμε ότι κάθε ευρώ που δαπανά μια ανθρωπιστική οργάνωση σε διαπεριτούς σκοπούς ουσιαστικά στερεί ένα ευρώ από τον εμβολιασμό των παιδιών ή από την παροχή γευμάτων σε παιδιά. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο να είμαστε όσο τον πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στη δραστηριοποίησή μας. Και οι ευρωβουλευτές ε, μας το επενθυμίζουν αυτό συνεχώς, αυτό είναι πολύ θετικό και μετά την ε, Σύνοδο κορυφή της Κωνσταντινούπολης είχαν γίνει μια σειρά δεσμεύσει που θα συμβάλλουν στην αύξηση τη αποτελεσματικότητας. Χρήση ρευστού που είναι αποτελεσματική σε μια σειρά περιπτώσεων, μακροπρόθεσμε δεσμεύσει, γιατί κάποιε από τι κρίσει που αντιμετωπίζουμε ε, διαιωνίζονται ή ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έτσι καλύτερο να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό παρά να αντιμετωπίζουμε κάθε φορά αποσπασματικά μια κρίση. Όταν ξεκίνησα στη θέση που ανέλαβα, ε, είπα στο επιτελείο μου το, τα 2.000 άτομα που εργάζονται στον Ότσα και κάνουν εξαιρετική δουλειά ε, σε εκατοντάδες σημεία του πλανήτη, ακόμα και σε μέρη της Συρίας που βαβαρδίζονται συνεχώς, και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με πολύ, σε πολύ δύσκολα σημεία και στη Σομαλία. Πραγματικά εξαιρετικό το προσωπικό μας, με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται. Ε, τους είπα λοιπόν ότι μέχρι το τέλος της θητείας μου θα ήθελα ο κόσμος να τα πηγαίνει καλύτερα σε ό,τι αφορά τρία βασικά προβλήματα. Πρώτον, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας προκύπτει από την ε, συμπεριφορά και την επιθετικότητα των ηθινόντων σε περιοχή συγκρούσεων και στη ε, Συρία και στην Ιεμένη και αλλού. Έχουμε δει ε, μία διολίστηση σε ό,τι αφορά την ε, τήρηση του διεθνούς δικαίου και αυτό οδηγεί σε επιθέσεις σε νοσοκομεία, σχολεία και ούτω καθεξής. Πρέπει κάτι να κάνουμε για να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Και στο παρελθόν είχαμε τέτοια προβλήματα και με στα Βαλκάνια στις αρχές του 1990 τραβούσαμε τα μαλλιά μας και λέγαμε πώ είναι δυνατόν θα υπάρξει ποτέ λογοδοσία. Και είδαμε ότι τελικά, ακόμα και αν αυτό πήρε πολύ καιρό, ο κύριος Μλάντιτς, ο κύριος Κάραντιτς και ο κύριος ε, Μιλόσεβιτς ε, ενώπιον της δικαιοσύνης στη Χάγη και δικάστηκαν. Ε, πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να επιμένουμε επί της σημασίας της ε, λογοδοσίας και της συλλογή ε, στοιχείων και μαρτυριών. Ο δεύτερος τομέας όπου θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος μέσα σε μερικά χρόνια έχει να κάνει με τις επιστημιστικές κρίσεις. Κατά τη γνώμη μου, ο λοιμός μπορεί να εξαλειφθεί. παλιότερα ήταν πανταχού παρόντες οι λοιμοί. Ε, και μάλιστα εγώ επειδή έχω και Ιρλανδική καταγωγή, από πολύ μικρός έμαθα για τον λοιμό της πατάτας ε, το 1840 που ένα εκατομμύριο Ιρλανδοί έχασαν τη ζωή τους και ένα εκατομμύριο μετανάστευσε. Αυτό συνέβαινε συνεχώς και παντού στον κόσμο. Τα τελευταία 50 χρόνια ο λοιμός έχει γίνει πολύ πιο σπάνιος και πολύ λιγότερο θανατηφόρος. Δεν υπάρχει ένας λόγος να μην εξαλείψουμε τον λοιμό γενικά από τον κόσμο και εξετάζουμε ορισμένες νέες πρωτοβουλίες για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Και ο τρίτος τομέας έχει να κάνει με τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες. Υπήρξε μία ισχυρή αύξηση ε, του προσφυγικού και εξαιτία της Συρίας, αλλά ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στους εκτοπιστέντες. Πολύ συχνά ο εκτοπισμός, δηλαδή όταν ε, ε, πολίτες μιας χώρας αναγκάζονται να αφήσουν το σημείο που μένουν και να πάνε σε άλλο σημείο της πατρίδας τους, ε, κάπως αφήνουμε να, να αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε λύσεις και μάλιστα γρήγορα και όχι να τους αφήνουμε να διαβιούν υπό απαράδεκτες ε, και ανθυγιεινές ε, συνθήκες τέτοιους καταβλισμούς. Πρέπει να έχουν δυνατότητα να χτίσουν τη ζωή τους και κάπου αλλού. Όπου έχω συνομιλήσει με πολλούς τέτοιους ανθρώπους και είπαν ότι αυτό που δεν θέλουμε τίποτα είναι να παραμείνουν στον καταβλισμό τους. Θέλουν να έχουν δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού. Ο ΙΕ φέτος προσπαθεί να θεσπίσει νέες πολιτικές που θα συμφωνηθούν από όλα τα κράτη-μέλη του ΙΕ για να αντιμετωπίσουν και προβλήματα των προσφύγων και της μετανάστευσης. Εάν τα καταφέρουμε σε αυτούς τους τρεις τομείς, μέχρι το τέλος της θητείας μου, θα θεωρώ ότι είχα μια επιτυχή θητεία. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο εδώ και να επαναλάβω, αν μου επιτρέπετε, το βασικό μου μήνυμα ότι η στήριξή σας προς εμάς είναι εξαιρετικά σημαντική και από τις αποφάσεις που λαμβάνετε ελπίζω να καταλαβαίνετε και τη διαφορά, ε, τη βοήθεια που παρέχετε σε εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Well, η πρόεδρος Μακάβαν. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε όχι μόνο ε, μια εικόνα αλλά και ιδέες για τη μελλοντική δουλειά μας. Έχετε ερωτήσεις εσείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ε, ε εσείς πρώτος. Πρώτα το Λαϊκό Κόμμα λοιπόν. Συμφωνώ πόσο ε, σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να έχουμε έτοιμη μια εύκαμπτη ατζέντα για να μπορούμε να αντιδρούμε με ταχύτητα. Για να είναι και η ανταπόκρισή μας πιο αποτελεσματική. Με αυτή την τελευταία έκθεση για την ασφάλεια διατροφής πρέπει να έχουμε του νου γιατί έχουμε ήδη κάποιες ε, προειδοποιήσεις για μετά το 2030. Έχουμε κάποιες επιτυχίες ως τώρα, αλλά πρέπει να δούμε και παραπέρα. Για την συλλογή δεδομένων, επειδή συζητούμε για την ψηφιοποίηση των δεδομένων, πώς βλέπετε τη δυνατότητα να ψηφιοποιηθεί η συλλογή δεδομένων για να βελτιωθεί η κατάσταση σε ορισμένες χώρες παραλήπτριες. Ας ακούσουμε πρώτα μερικές απόψεις, ερωτήσεις και μετά μπορείτε να απαντήσετε. Εσείς θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάπτυξη του θέματος που βασίζεται βέβαια σε πολύχρονη εμπειρία. Είναι σημαντικό να το επαναλάβω με αυτό. Αρχικά μας είπατε πολλά θετικά νέα. Ξεκολουθούμε να είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές η αποτελεσματικότητα έχει βελτιωθεί. Είπατε επίσης ότι παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί να είναι αναγκαίο να απορροφώνται πολλά χρήματα σε μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ ως Ευρωκοινοβούλιο, επειδή πρέπει Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπερασπιστούμε τον προϋπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, ο οποίος δέχεται συνεχώς επιθέσεις. Η κατάχρηση των κονδυλίων αυτών μάλλον πάνε να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς σκοπούς μέσα στην αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά όχι η ανθρωπιστική βοήθεια. η, αναπτυξιακή, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραμείνει καθαρά ανθρωπιστική βοήθεια. Από την άλλη μεριά έχουμε δικαίωμα να είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι εξακολουθούμε να είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές. Και ότι η αποδοτικότητα της βοήθειας αυτής έχει προχωρήσει κι άλλο και δεν καλύπτουμε πια μόνο τις καθημερινές ανάγκες, αλλά και ιδίω μιλούμε για την βοήθεια σε πρόσφυγες και σε εκτοπισμένους. Νομίζω αυτό που ανέφερε πριν ο συνάδελφός μου Bogdan Μένσον είναι ότι πρέπει να δούμε και την ευθύνη. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί μέσα εθνικές κοινότητες, όχι μόνο όπως στη Σερβία, αλλά πρέπει να βάλουμε μυαλό και η διεθνής κοινότητα δηλαδή να αντιληφθεί ότι Εάν υπάρχουν ευθύνες, αυτές πρέπει να αποδίδονται. Άλλωστε είμαστε υπεύθυνοι και απέναντι, υπόλογοι δηλαδή, απέναντι στους φορολογουμένους, οι οποίοι μας απαιτούν από εμά αυτή την αποτελεσματικότητα. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν και κατέθεσε μια καλή ιδέα, να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε κοινότητες όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα προσφύγων. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν, α, ε, δεν επαρκεί η αλληλεγγύη από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ορισμένες χώρες όπως ε, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία δεν δείχνουν το ίδιο επίπεδο αλληλεγγύη. Ε, να επενδύουμε χρήματα στις περιφέρειες και στις τοπικές εκείνες αρχές που επιθυμούν να βοηθήσουν πρόσφυγες. Να μην προσπαθήσουμε αναγκαία να επιβάλλουμε με κυρώσεις σε άλλους που δεν δείχνουν την αλληλεγγύη αυτή, αλλά να βοηθήσουμε ιδιαίτερα αυτούς που δείχνουν. Και πέραν τώρα από το ότι είμαστε μεγαλύτεροι δωρητές, τι γίνεται με χώρες άλλες σημαντικές, με σημαντικές αναπτυγμένες οικονομίες όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Ινδία. Ποιος είναι ο ρόλος τους στην στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας. My two colleagues, so we'll take those first, then see if any other. I've got a couple of points I want to ask. Πολλές ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις ε, και ε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικές οι ερωτήσεις σας για τον κύριο Φέντερς να πω. Πιστεύω ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει μία ευκαιρία μεταμόρφωσης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για να προβλέψουμε τα προβλήματα που μάλλον θα συμβούν και να ενεργήσουμε νωρίτερα, ε, πιο έγκαιρα. Δηλαδή, όχι μόνο το να μειώσουμε τα προβλήματα, αλλά είναι και πολύ φθηνότερο το να μπορούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα. Κοστίζει πολύ λιγότερο. Επίσης, εργαζόμαστε σε ένα φάσμα νέων τρόπων για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στα στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να ενεργήσουμε νωρίτερα. Ε, να σας κάνω ένα παραλληλισμό. Στις είπα, όταν οι αρχές για τη δημόσια υγεία ε, κάνουν μία σφιγμομέτρηση και προσπαθούν να δουν ή να εξετάσουν πώς θα, ε, πότε θα υπάρξει η να εξετασουν πως επιδημία γρήπης βλέπουν ε, τον αριθμό των ανθρώπων που επισκέπτονται στο το γιατρό και τον αριθμό των ανθρώπων που επισκέπτονται το φαρμακείο τους, αλλά βλέπουν επίσης ε, πολύ κόσμο που κοιτάει στα iPad ή στα κομπιούτερ και ψάχνει να δει ποια είναι τα συμπτώματα της γρήπης. Ε, υπάρχει πολύ έντονη συσχέτιση μεταξύ αυτής της παρατήρησης και της επόμενης επιδημίας να σας πω ας πούμε ότι στη Σομαλία στις αρχές του, του περασμένου χρόνου η χρήση των στοιχείων στα κινητά τηλέφωνα μειώθηκε γιατί εξαντλούσαν τους πόρους τους και αυτό ήταν ένας, ε, μια ένδειξη ότι ο κόσμος ήταν πολύ ευάλωτος σε λοιμό. Αυτό το ίδιο οι τεχνικές είναι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι το πρώτο μου παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα είναι η χρήση του blockchain και των κινούμενων χρηματών για να μπορέσουμε να βρούμε ε, και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ο μεγαλύτερος λόγος που έχασε τη ζωή του από λοιμό στη 1,5 εκατομμύριο κόσμο στη Σομαλία ήταν γιατί η Al-Shabaab ε, μπόρεσε να περιορίσει και να επιβάλλει το νόμο στις ε, περιοχές που ήλεγχε είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορέσει κανείς να κρατήσει όμοιρο ε, το blockchain ή το mobile money από ότι να ε, εμποδίσει, να περιορίσει την αποστολή επιστησικής βοήθειας στις περιοχές που ελέγχει. Μάθαμε λοιπόν από την περασμένη χρονιά ότι ας πούμε με μηνύματα και με τα κινητά τηλέφωνα ε, το σύστημα αυτό λειτουργεί. Ακόμα και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα το να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακή τεχνολογία βοηθά τον κόσμο, πράγμα που δεν το είχαμε στο παρελθόν. Θα μπορούσα να σας μιλάω άλλη μισή ώρα γι' αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που με συναρπάζει, είναι μια τεράστια ευκαιρία για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και λειτουργούμε. Στις δικέ σα ερωτήσεις τώρα κύριε Νόρφοκ, να πω ότι τα ζητήματα που θίξατε είναι ακριβώς αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τον Επίτροπο Στυλιανίδη, του συναδέλφου στην ΕΚΟ, στις συζητήσεις που έχουμε μαζί τους. Ελπίζω πως ε, το Ευρωκοινοβούλιο είναι περήφανο για το ρόλο που παίζει η ΕΚΟ. Είναι μια από τις πιο καλές ανθρωπιστικές υπηρεσίες στον κόσμο. Κάνουν υπέροχη δουλειά. Ελπίζω να καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο, ε, πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη της ΕΚΟ για την Ευρώπη. Η ανθρωπιστική δράση είναι ένας πολύ φθηνός τρόπος για να σωθούν ε, ζωές. Κοστίζει περίπου 70 cents την ημέρα για να σωθεί η ζωή κάποιου που έχει ε, παγιδευτεί σε μια ανθρωπιστική κρίση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα και πριν, οι υπηρεσίες βοήθειας να χρησιμοποιηθούν καλά τα χρήματά τους. Εγώ είμαι λογιστής ε, αρχικά, ε, μετά σπούδασα οικονομικά και ε, business. Ποτέ όμως δεν αρκούν τα χρήματα, γι' αυτό πρέπει να βρούμε τους καλύτερους τρόπους πάντα να τα διαχειριστούμε και αν δεν τα διαχειριστούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τότε δεν σώζουμε όσους θα μπορούσαμε να σώσουμε. Επίσης σημαντικό είναι ότι τα δύο τρίτα των χρημάτων που έχει ετησίως ο ΙΕ ε, για ανθρωπιστική βοήθεια προέρχεται από τους πέντε κύριους δωρητές και αυτός ο αριθμός, αυτό το μερίδιο θα πρέπει να διευρυνθεί με τις κυβερνήσεις της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συζητήσαμε μια συμφωνία 190 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ιεμένη. Η μεγαλύτερη βοήθεια ε, που έχει υπάρξει ποτέ σε μια μόνη πληρωμή δόθηκαν όλα αυτά τα χρήματα. Είναι στην τράπεζα του ΟΗΑ αυτή τη στιγμή τα χρήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερα ε, παραδείγματα ώστε ο κόσμος που μπορεί να συμβάλλει περισσότερο να το κάνει και να παίξει πιο σημαντικό ρόλο και ελπίζω πως θα σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό τα επόμενα χρόνια γιατί είναι εύκολο και είναι προς το συμφέρον όλων τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπίζονται. Τώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο είναι καλύτερο τα προβλήματα να διορθώνονται εκεί που εκδηλώνονται και να μην ε, τους επιτρέπεται να εξαπλωθούν. Όλοι θυμόμαστε πως το 2015 ένα εκατομμύριο κόσμος ήρθε στην Ευρώπη κυρίως από τη Συρία και αυτό εν μέρη διότι η προσπάθεια που καταβάλαμε το 2014 για να καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου αυτού εκεί που βρισκόταν δεν ήταν επιτυχής από ό,τι ήταν και λιγότερο επιτυχής από ό,τι το 2012 ή το 2013. Όποια μηνύματα που θέλω να διαβιβάσω αυτή την εβδομάδα είναι ότι είναι σημαντικό να χρηματοδοτηθεί σωστά η δραστηριότητά μας, να έχουμε αρκετούς πόρους, πρώτη προτεραιότητα είναι για την Ιορδανία, το Λίβανο και την Τουρκία που είναι, ε, φιλοξενούν το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, ώστε να τους φροντίσουν, αλλά και να διατηρηθεί η σταθερότητα, κυρίως του Λιβάνου και της Ιορδανίας, που έχουν αναλάβει τεράστιο βάρος τα τελευταία χρόνια. Όλα τα προβλήματα πάντως είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται εκεί όπου εκδηλώνονται και όχι να πρέπει να αντιμετωπιστούν αργότερα και σε πολύ περισσότερα μέρη. Ο Νόρμπερτ και εγώ επισκεφθήκαμε καταβλισμού προσφύγων στην Τουρκία το Σεπτέμβριο του 2015 και ήμασταν εκεί ακριβώ τότε που εξεράγει όλη αυτή η υπόθεση. Εγώ αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι ο θυμός των τουρκικών αρχών που αισθάνονταν ότι έχουν μείνει μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τα πάντα. Και αυτή η οργή μετατράπηκε στο εντάξει τότε θα ανοίξουμε τις ε, πόρτες και τότε θα δείτε τι θα γίνει αν δεν μας βοηθήσετε να χρηματοδοτήσετε αυτή την κατάσταση. Είναι καλό να το θυμίζουμε αυτό γιατί αργότερα στην συνεδρίασή μας έχουμε ερωτήσεις προς την Επιτροπή και μια από τις ερωτήσεις που ένας συνάδελφος θα υποβάλει αφορά την διάσκεψη για τη Συρία αυτή την εβδομάδα και λέει ότι από την έκκληση του 2017 για τη Συρία μόνο το 50% έχει βρεθεί και μόνο το 40% έχει δοθεί στην πράξη. Μέχρι πέσιο το 53% λοιπόν είχε χρηματοδοτηθεί από τις ανάγκες και μόνο 30 δις έχουν δεσμεύσει οι δορυτές. Δηλαδή πολλοί λένε ότι θα δώσουν αλλά στην πράξη ε, δεν το κάνουν. Δεύτερη παρατήρηση. Και με χαρά άκουσα τα όσα είπατε για ολόκληρη την υπόθεση της συμμόρφωσης προς ε, το διεθνή, ανθρωπιστικό, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ότι δηλαδή θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε να γίνονται σεβαστε, γίνεται σεβαστό το δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο. Στο γραφείο Ζαχάροφ δόθηκε σε δύο γυναίκες σε Γεζίδι που, από το Ιράκ και μια από εκείνες ε, κατονόμασε το Γενικό Διευθυντή ενός νοσοκομείου στην ε, πόλη της που την είχε ε, καταχραστεί. Και τότε ρωτήσαμε την Κομισιόν, θα αντιμετωπίσετε όχι μόνο την ανθρωπιστική κατάσταση, αλλά και όλες αυτές τις καταχρήσεις και τις ε, ο κόσμος να δει δηλαδή ποια είναι η συνέπεια όταν έχεις τέτοια συμπεριφορά. Ένοπλες συγκρούσεις, ε, χαοτικές καταστάσεις, ε, οι κυβερνήσεις που δεν δικάζονται από το Διεθνές Δικαστήριο. Τώρα μου αρέσει η ιδέα της κρίζωσης της πείνας στο PDP ε, για τον προπολογισμό 2021 μέχρι 2027 έχουμε μια ολόκληρη γενιά προγραμμάτων. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαν οι συνάδελφοι που θα είναι εδώ τον, στην επόμενη θητεία να, αν η εκρίζωση της πείνας θα είναι ε, στόχος. Εσείς ξέρετε τα, τα, τα, ποια είναι τα δικά μας ε, μέσα. Έχετε εργαστεί στο DFID. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει εκεί. Και τέλος, για τους πρόσφυγες, τους εκτοπισμένους, εσωτερικά εκτοπισμένους, κυρίως στις γειτονικές χώρες, ποια είναι τα καλύτερα παραδείγματα από αυτά που έχετε δει για το πώς ε, αντιμετώπισαν οι χώρες τους εκτοπισμένους ε, υπάρχουν διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε. Πάμε στην Ουγκάντα. Μου λένε ότι είναι καλό παράδειγμα η Ουγκάντα γιατί δίνει τη δυνατότητα στους πρόσφυγες ε, να καλλιεργήσουν ε, γη και να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Και στην Τουρκία είδαμε εντυπωσιακά παραδείγματα προσπαθειών της τουρκικής κυβέρνησης να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Έχουν μια αγορά, έχουν σούπερ μάρκετ, ε, ε, μπορούν να χρησιμοποιούν κάτι κάρτες που έχουν φτιάξει για να ανταλλάσσουν ε, τρόφιμα. Να έχουν μια πιο φυσιολογική οικογενειακή ζωή δηλαδή. Αυτά έχω να πω. Κάποιο από του συναδέλφου μόλι έφτασε, ο κύριο Σαφχάουζερ, και θέλει και εκείνο να θέσει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, έχουμε και την Επιτροπή Άφετ και εγώ πήρα το λόγο για τη Λιβύη και δεν μπορούσα να μεταφτώ χρόνο και στις δύο. Ο βοηθός μου όμως με ενημέρωσε για τη συζήτηση που γίνεται. Έχω μια ερώτηση Καταρχάς δεν πιστεύω πως το σύστημα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Το λέω α, με βάση μια εμπειρία. Δεν λέω το δικό μας σύστημα, αλλά λέω γενικότερα το σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας. Και γιατί το λέω, γιατί διαπιστώνουμε συστηματικά, παρατηρούμε συστηματικά την καταστροφή κρατών, όπως στη Λιβύη ας πούμε. Μετά το ίδιο θα είχε γίνει και στη Συρία αν δεν είχαμε μπορέσει χάρη στη Ρωσία να σώσουμε τον Ασάντ. Και σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει πλέον κράτος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αποτελεσματική κατανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Περνάμε από τις ΜΚΟ, αλλά αυτό που είναι βέβαιο, και εδώ θέλω να σας θέσω και την ερώτησή μου, ότι αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αν δούμε τις ΜΚΟ, και αν συνεχίσουμε να πυρνάμε μέσα από αυτό, έχουμε μέγα μέλλον. Ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο μόνος τρόπος ε, για να υπάρξει ανάπτυξη ε, είναι ένα κράτος να αναλάβει την ίδια του την ανάπτυξη. Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Ποτέ δεν είδαμε μια μη κυβερνητική οργάνωση να μπορέσει να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της χώρας. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή όπου εμείς βοηθάμε μόνο τις ΜΚΟ να βοηθήσουν επιγόντως, πέφτουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Και μπορώ να σας πω ότι ναι, εσείς παρεμβαίνετε, θα παρεμβαίνετε και ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, μέχρι ότου δεν θα υπάρχουν πια χρήματα. Γιατί παντού θα συμβαίνει το ίδιο. Εσείς πώς βλέπετε να μπορούμε να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Η ερώτηση που σας έτω δεν αφορά το δικό σας επάγγελμα, ε, αλλά πώς βγαίνουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Καλούμεθα να βοηθήσουμε, θα στο μέλλον να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο και αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν πρόκειται να αποκαταστήσουν την ανάπτυξη και δεν θα βοηθήσουν να παρεμβαίνουμε λιγότερο. Πώς θα βγούμε από τον φαύλο κύκλο, Πώς θα αποκαταστήσουμε και θα ξανασυστήσουμε κράτη. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα επί του οποίου θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Ακούσατε πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για απάντηση. Να αρχίσω με την ερώτηση που κάνατε για τη Συρία. Δεν γνωρίζουμε πώς θα χρηματοδοτηθεί η έκκληση που κάνουμε φέτος ζητούμε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες 13 εκατομμυρίων σύρων μέσα στην ίδια τη χώρα, 4,5 δισεκατομμύρια για την ανταπόκριση της ανάγκης των προσφύγων εκτός χώρας. Μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι θα γνωρίζω την απάντηση στην ερώτησή σας και θα τη διοχετεύσω στον τύπο. Αλλά, όπως είπα, Καλά θα κάνει ο κόσμος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να φανεί γενναιόδωρος. Γιατί είδαμε το 2015 τι έγινε όταν η απάντηση ήταν λιγότερο γενναιόδωρη. Τι μπορούν να κάνουν συλλογικά τα ευρωπαϊκά όργανα για να συμβάλλουν περισσότερο στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της απάλληψης της πείνας και για να υπάρξει ασφάλεια διατροφής. Χρειάζεται μια όσο γίνεται πιο μακροπρόθεσμη προοπτική στην, ε, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Πολλά πράγματα από αυτά που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό ΑΚΕ που έχετε. Υπάρχουν λοιπόν σχετικά παραδείγματα. Και είναι σωστό το μοντέλο που ακολουθείτε. Μακροπρόθεσμα δηλαδή. Όσο περισσότεροι λειτουργήσουν το ίδιο και μπορέσουμε να βάλουμε μαζί αυτέ τι 30-40 χώρε. να συμπορευτούν, αλλά να είμαστε και ρεαλιστέ. Διότι ορισμένε χώρε, οι οποίε είναι ευάλωτε σε ξηρασίε, θα αντιμετωπίσουν περισσότερε και μακρότερε περιόδου ξηρασία λόγω τη αλλαγή του κλίματο. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να γίνει, εκτός από την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους, είναι να φτιάξουμε αποτελεσματικά δίκτυα ασφαλείας τα οποία να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά μόλις προκύψει το επόμενο πρόβλημα. Και αυτός είναι και ο πιο οικονομικός τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς τα προβλήματα αυτά σε χώρες που πλήττονται από ξηρασία. Μακροπρόθεσμες λύσεις στην ε, επισφάλεια διατροφής είναι τα ίδια περίπου. Είναι πολιτικά συστήματα τα οποία πρέπει, οφείλουν να αποκρίνονται τις ανάγκες των ε, κατοίκων και ανάπτυξη. Δεν υπάρχει βέβαια μια συνταγή που να τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Χώρες που τα έχουν πάει καλά τα τελευταία 15 χρόνια είναι ότι είναι αυτές που έχουν πορευθεί κατάλληλα και στα τρία αυτά. Για τους εκτοπισμένους και για επιτυχή παραδείγματα Υπάρχουν τέτοια. Μπορούν, κάποιες χώρες έχουν βοηθήσει τους εκτοπισμένους να έχουν πρόσβαση σε γη και σε τρόπο να ξαναβάλουν μπρος οικονομικά τη ζωή τους. Και στη διάσκεψη του Λονδίνου το 2016 σε ένα σύμφωνο, έγινε ένα σύμφωνο για να στηριχθεί η Ιορδανία να επιτρέψει περισσότερα νεαρά σιρόπουλα να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα και να δώσει και άδειε εργασία ώστε Σύριοι να μπορέσουν να εργαστούν πολύ καλύτερη προσέγγιση αυτή για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους προσφυγικές κρίσεις από το να κρατάτε τον κόσμο σε μεγάλα κέντρα ε, προσφύγων. Η εμπειρία από το 2016 και μετά είναι αρκετά θετική. Και τα ίδια, ίδια είδαμε και στο Λίβανο και στην Αιθιοπία. Για την τελευταία ερώτηση που μου έκανε ο συνάδελφός σας, όπως είπα προηγουμένως, δουλεύω παραπάνω από 30 χρόνια στα πράγματα αυτά. Το σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας έχει διασώσει εκατομμύρια ανθρώπους και διασώζει κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ότι βεβαίω θα ήταν καλύτερα να μην συνέβαιναν τα πράγματα αυτά. Κανείς δεν θέλει να βλέπει να χάνονται μαζικά ζωές ανθρώπων. Προφανώς τα διάφορα κράτη πρέπει να παίζουν τον θεμελιώδη ρόλο σε κάθε χώρα μέσα για να δημιουργούν τις συνθήκες ε, να μπορούν να ζήσουν και να επιζήσουν οι πολίτες τους. Σε ορισμένε περιπτώσεις όμως το συγκεκριμένο κράτος δεν είναι διατεθειμένο ή δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Και γι' αυτό σε ψήφισμά του το Συμβούλιο Ασφαλείας το 1991, με το οποίο δημιούργησε και τη θέση την οποία κατέχω, συμφώνησε ότι εάν ένα κράτος δεν είναι διατεθειμένο ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τότε παρεμβαίνει η διεθνή κοινότητα και συχνά οι μη κρατικέ οργανώσεις κάνουν καταπληκτική δουλειά στο τελευταίο μέρος του συστήματος υλοποίηση των ε, στόχων του συστήματος ανθρωπιστικής βοήθειας, διότι γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα επιτόπου. Οι μη κρατικές οργανώσεις και κατά τη δική μου εμπειρία σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες παίζουν σημαντικότατο ρόλο και σε άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών και ιδίως στην λογοδοσία των υπευθύνων των κυβερνήσεων. Σε όλες τις χώρες μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις διαφόρων ειδών μεταξύ αυτών ο τύπος, ομάδες λόμπι, παρόχων υπηρεσιών παίζουν θεμελιώδη ρόλο στην πολιτική ζωή. Οι NGO λοιπόν δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το κράτος, αλλά σε κάθε κράτος, είτε είναι αναπτυγμένο, είτε βρίσκεται σε κρίση ή κάπου ενδιάμεσα, οι ε, μη κρατικέ οργανώσεις έχουν, θεωρώ, θεμελιώδη ρόλο να παίξουν. Άλλο θέμα είναι αυτό που έχουμε συζητήσει και που είναι ο πολύ συμπιεσμένος χώρος για να αναπτύξουν δραστηριότητες οι, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Βεβαίω ο ρόλο του δεν είναι να επενούν τι κυβερνήσει, είτε αυτέ που είναι σε Βρυξέλλε, είτε αυτέ που είναι σε διάφορε χώρε. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ, Μάρκ, και μα δώσατε πολύ τροφή για σκέψη, καθώ αναπτύσσουμε τον νέο σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο. Αν έχετε και άλλε σκέψει για την ανθρωπιστική βοήθεια και για την αναδιάρθρωσή της. Άλλωστε ε, συνεργαζόμαστε στενά με τον Επίτροπο Στυλιανίδη και συμμεριζόμαστε τη δέσμευσή του για την προστασία των προσφύγων και ελπίζω ε, να είναι επιτυχία η διασκεψή σας και όχι μόνο να ε, αναλάβουν δεσμεύσεις οι υπεύθυνοι αλλά και να σας διαθέσουν όντως τη χρηματοδότηση που ζητείτε. Uh, Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 7. Προπολογισμό. Είπαμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τον ε, προπολογισμό ε, και κάτι καταφέραμε μάλλον πέρυσι να το κάνουμε αυτό, να μην περικοπεί ο ε, προπολογισμό για την ανθρωπιστική βάση. Τώρα θα συζητήσουμε το 2019 και με τον ε, Γενικό Εισηγητή κύριο Ντανιέλε Βιώτη. Θα σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Περιμένατε και μερικά λεπτά, αλλά καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ σημαντικός ο καλεσμένος μας. Ελπίζουμε να έχετε καλά νέα για μας για το 2019. Παρακαλώ, αυτή το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου αναθέτεται αμέσως μια μεγάλη ευθύνη να δώσω καλά νέα για σήμερα. Δυστυχώς δεν είμαι ακόμα σε θέση σήμερα βεβαίως. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για αυτήν την ε, σημερινή συνάντηση που σίγουρα θα είναι, ε, πολύ χρήσιμη. Καταρχάς, ε, να σας πω μια, κάτι για την μέθοδο. Πρόθεσή μου ως εισηγητής για τον προπολογισμό του επόμενου χρόνου είναι να έχω όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή και μεγαλύτερη... συνεργασία για τη δουλειά που θα γίνει στη διάρκεια της τελικής ε, συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και γι' αυτό και ξεκινάμε από σήμερα σε συνεργασία με την, και με τη δική σας Επιτροπή. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στα κύρια σημεία που φαντάζομαι ενδιαφέρον την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, και που ήδη περιλαμβάνονται μέρη στην δράση στις κατευθυντήριες γραμμές που ψηφίσαμε τον Μάρτιο και που θα αποτελέσουν τα κεντρικά σημεία για το προπολογισμό του επόμενου έτους. Καταρχάς, ε, η πάντοτε ε, πολύ έντονη σκέψη και προσοχή στο φαινόμενο των μεταναστών, των προσφύγων και των ετούντων άσυλο. προσοχή και λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε τις δαπάνες και τις εξελίξεις με βάση τις διάφορες κρίσεις που μπορεί να προκύψουν πέρα από τον ε, προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κληθεί να δώσει περισσότερη ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Έπειτα ε, το θέμα των προσφύγων στην Τουρκία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα όπως γνωρίζετε θα έπρεπε να ξεκινήσει η χρηματοδότηση του δεύτερου τμήματος της διευκόλυνση για την Τουρκία, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μέσα στο Συμβούλιο για το πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Η Κομισιόν πρότεινε να συνεχιστεί και εμείς συμφωνούμε ε, με αυτό, να συνεχιστεί αυτό που έγινε με το πρώτο τμήμα ε, ε, συμβολή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών Ακόμα δεν έχει υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες χώρες στο Συμβούλιο που θα ήθελαν να αφήσουν το σύνολο των 3 εκατομμυρίων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια αυτό για μας δεν είναι αποδεκτό ως θέση ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους. Θα δούμε έπειτα τι θα συμβεί ε, μεθαύριο με την ε, διάσκεψη για τη Συρία που θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες. Επ' αυτό έχουμε ήδη δεσμευθεί ε, με ένα 1,275 δις για το 2017 και ελπίζουμε πως θα επιβεβαιωθούν και τα 560 εκατομμύρια για το 2018 με 2020. Πολύ σημαντικό επίσης για σας και για ολόκληρο το Κοινοβούλιο πιστεύω, για όλους, για όλους μας, είναι το θέμα που αφορά το Urban. δηλαδή την υπηρεσία του ΟΗΕ για την απασχόληση των Παλαιστινίων προσφύγων. Αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τους επόμενους μήνες ε, τις συζητήσεις γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την απόφαση των ΙΠΑ <coughs> να αρνηθούν την παραδοσιακή του συμβολή σε αυτή την υπηρεσία, σε αυτόν τον οργανισμό. Κάπως ε, θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το, το, ποσό, θα συνομιλήσουμε με την Ούρμπα, ε, ίσως θα υπάρξει κάποια δέσμευση από πλευράς μας. Τέλος, δύο τελευταίες ε, σκέψεις για τις ανθρωπιστικές δαπάνες, για τις δυσμεύσεις και τις πληρωμές που και σε αυτή την περίπτωση θα είναι προτεραιότητας γιατί προέρχονται όλες αυτές, όλες αυτές τις ανάγκες από την αύξηση των προσφύγων. Μιλώ για το σύνολο των ε, ένοπλων ε, συγκρούσεων στην Συρία, στην Ιεμένη, στο Ιράκ, στην Ουκρανία, το Αφγανιστάν, τη Μιανμάρ, τη Λιβύη, Τσάντ, κέρας της Αφρικής, ε, καθώς και τη σταδιακή αύξηση της συχνότητας των φυσικών καταστροφών και λόγω των κλιματικών αλλαγών. Πολύ σημαντικό επίσης θέμα το του πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας. στο σημείο το πιο σημαντικό που Ε, στηρίζει τη θέση της Επιτροπής ε, ΔΕΒΕ είναι ότι τόσο το ε, μέσο αναπτυξιακής βοήθειας όσο και η ανθρωπιστική βοήθεια όπου υπάρχει ε, πολύ μεγάλη, πολύ καλό επίπεδο δεσμεύσεων και υποχρεώσεων και πληρωμών. Και εδώ ε, νομίζω πως αυτό μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Thank you, thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι εδώ η Ανιλίνης που είναι η συζητητρία για αυτή τη δική μας ομοδότηση, αλλά Νόρπερτ παίρνει το λόγο να και την εκπροσωπείς ναι, αλλά νομίζω ότι ο συνάδελφο Ρούμπικ είναι εισηγητή και η Άννα Λίτ είναι σκιώδη. Μπορώ όμω να εκπροσωπήσω τη σκιώδη. Όχι, Άννα είναι εισηγητρία. Έχω ορισμένε παρατηρήσει. Δεν έχει σημασία αν είναι του, σκι... του εισηγητή ή του σκιώδου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Ντανιέλε. από την Επιτροπή Προπολογισμών. Υπάρχουν ορισμένε προτεραιότητε για τον προπολογισμό του 19 που θα ήθελα να αναφέρω. και τις οποίες θα θίξουμε και στην γνωμοδότηση. Εν γέννη, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να συνάδει με την εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να επενδύσουμε στην παιδεία, ε, να ενισχύσουμε τις ε, γυναίκες και τα παιδιά ε, και δράσεις κατά πολέμηση κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ή αναμένουμε τουλάχιστον μια διατήρηση των πιστώσεων ανάλυση χρεώσεων και πληρωμών στο TCI. Ένα σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι δεν θα υπάρξουν κονδύλια TCI προς την ασφάλεια και ειρήνη, όπως είχε συμφωνηθεί στους τριμερείς διαλόγους για τις ε, τροπολογίες ως προς αυτό το χρηματοδοτικό μέσο. Επιπλέον πρέπει να διατηρήσουμε την έμφαση στη μετανάστευση και να μην υπάρξουν περικοπές στις συνεισφορές του 19. Παράλληλα, προτεραιότητα είναι η παροχή πραγματικής ανθρωπιστικής βοήθειας, για να υπάρχει ποιοτική και συνεκτική ανθρωπιστική βοήθεια. Ζητούμε λοιπόν την αύξηση των πληρωμών σε αυτούς τους δύο τομείς. Προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος ε, βιώσιμης ανάπτυξης ε, υπαριθμών 13 προβλέπει την ανάληψη δράσης ε, για το κλίμα. Χρειάζεται λοιπόν σχετική διπλωματία και προσαρμογή του προπολογισμού στον τίτλο 4, τομέα 4. Ε, αυτά από την Άννα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Χάουτελε. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Ακόμα και αν αυτή η συζήτηση γίνεται χωρί έγγραφα, γιατί είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την προβολή του 19, θα ήθελα να επισημάνω τι πρόσφατε επιφυλάξει ε, που εξέφρασαν αρκετοί στην ενδιάμεση αναθεώρηση του EDF και του TCI, που ευνοούσαν τη χρηματοδότηση για τον ιδιωτικό τομέα, τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Και όλα αυτά σε βάρος ε, Παραδοσιακή ανθρωπιστική ανάπτυξη, δηλαδή κονδύλια για την ε, υγεία και την παιδεία. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ακόμα χρειαζόμαστε ισχυρέ ενέργειες για την ανθρωπιστική βοήθεια και ανάπτυξη. Να επισημάνω επίσης ότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες δημόσιες διαπάνες και εκεί η γραμμή προλογισμού έχει περιοριστεί στον φετινό προπολογισμό. Αμέριστη είναι, η στήριξή αμέριστη είναι η στήριξή μου προς την κοινωνία των πολιτών και ε, τη στήριξη των ε, τοπικών αρχών στην ανάπτυξη. Κατάλληλη χρηματοδότηση χρειάζεται και για την ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί έχουμε τόσες διαφορετικές κρίσεις αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων Συρία, Νότιο Σουδάν, Ουκρανία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το καθεξής. Ευχαριστούμε. Και κ. Βέντα. Και ως Πολωνός, αλλά γενικά και ως μέλος της Επιτροπής πρέπει να ε, αναφέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το στοιχείο. Η ομάδα μας θα στηρίξει αυτή τη θέση και συμφωνώ και ορμισμένες από τις παρατηρήσεις. Πρέπει να εμπλακούν και οι μικρές επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στηρίζουμε αυτή τη θέση. Πράγματι θα είναι θετικό εάν μιλήσουμε για την ευθύνη για το σύνολο του προπολογισμού 19. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο. Ένα ερώτημα έχω εγώ με βάση τα όσα είπαν οι προηγούμενοι μιλητές για την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Κάναμε τις ε, Δεσμεύσει αυτέ στη συνδιάσκεψη των Παρισίων και κανονικά θα πρέπει τώρα να αρχίσουν οι πληρωμέ. Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ έλεγε ότι προσωπικά έχει δώσει τα ποσά που θα πρέπει να δώσουν οι Ηνωμένες η ελλείψη ε, χρηματοδότησης. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται ότι θα κάνουν αυτέ τι πληρωμέ. Αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τον προβλέψιμο του 19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντανιάλ Νταμίκο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπω ξέρετε, το Σώμα των Επιτρόπων δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το προσχέδιο προπολογισμού του 19. επομένω, ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για να σα παρουσιάσουμε. Από πλευρά μα έχουμε σημειώσει με μεγάλη προσοχή τις ε, προτεραιότητες των μελών της Επιτροπής και ιδιαίτερως εκτιμούμε και την εισαγωγή του εισηγητή ελπίζουμε να υπάρξει αγαστή συνεργασία μεταξύ μας. Σε αυτή τη φάση μπορώ μόνο να σας πω ότι γενικά συμφωνούμε με τις προτεραιότητες που έχετε επισημάνει και ιδίως ό,τι αφορά το DCI την ανθρωπιστική βοήθεια. Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι υπάρχει υψηλό συντελεστή εκτέλεση Είναι βασικό σημείο που πρέπει να εξετάσουμε και να βασιστούμε και για τη συζήτηση για την επόμενη χρονιά, γιατί φαίνεται ότι τα δύο αυτά μέσα έχουν θετικά αποτελέσματα, τουλάχιστον σε ποσοτικά στοιχεία, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι αντίστοιχη και ποιοτική εικόνα. Έχουμε σημειώσει λοιπόν όλες ε, τις ε, προτεραιότητες που έχετε εκφράσει σε αδρές γραμμές. Ελπίζουμε να υπάρξει καλή συνεργασία και βεβαίως είμαστε τεθειμένοι να συζητήσουμε σε όλη τη διάρκεια της ε, διαδικασίας τυχόν εκρεμή ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ακόμα νωρί λοιπόν. Τα θέματα είναι επιτάπητο. Ο εισηγητή και πάλι. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για τις παρεμβάσεις τους που είναι ήδη πολύ πολύ χρήσιμες από τώρα και έπειτα βεβαίως θα γίνει ακόμα πιο πολύτιμη η συνεργασία στις επόμενες φάσεις. Έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με τον συνάδελφο Πόλο Ρούμπλικ που είναι ο συνάδελφος στην Επιτροπή Προπολογισμού μαζί με εμένα ε, και σίγουρα θα έχουμε την δυνατότητα να συντονιστούμε γιατί η μόνη ερώτηση που επιβάλλατε εσείς Πρόεδρε για τις κλιματικές αλλαγές και τη Συμφωνία του Παρισιού δεν μπορώ να απαντήσω ακόμα ίσως αύριο να έχουμε γιατί αύριο έχουμε μια ακρόαση με την Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό για την ε, ρόλο του προϋπολογισμού και της σύμβασης του Παρισιού. Οπότε αύριο θα μπορώ να σας απαντήσω με περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, αυτό. Είναι πολύ θετικό που η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού ήδη συζητά τα θέματα. Όπως είπαμε ήταν η πρώτη φορά, δεν έχουμε έγγραφα. The lead... Uh, no, the, the, when what's the time? I'm looking at the timetable. So the Commission will present its draft budget on the... Η Κομισιόν θα υποβάλει το σχέδιο προπολογισμού 23 Μαΐου και εμείς θα αντιδράσουμε υπό τη μορφή επιστολών. Μάλιστα και στη συνέχεια θα συνταχθεί και επίσημο γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά το να φτιάξει τον προπολογισμό. Το ξέρουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν για όσα κάνει. Ευχαριστούμε και πάμε στο. Φεύγουμε από το 7 και περνάμε σε ένα νέο σημείο 8 που είναι το παλιό σημείο 21 πρώην 21 8. Αρχίσαμε ε, συμφωνώντας ε, ότι θα γινόταν αυτή η αλλαγή στην ημερήσια, ώστε αντί να ακούσουμε το, να συζητήσουμε μάλλον το 8, να συζητήσουμε το 21 τώρα. Ε, ενώ και Ιράκ. Εταιρική σχέση και συνεργασία. Το έχουμε ξαναδεί. Το 2013 το Κοινοβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας εταιρική σχέση και συνεργασίας με το Ιράκ. Μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την νομική βάση αυτής της συμφωνίας, παρόμοιε απόφασει, μάλλον με τι Φιλιππίνε, το Συμβούλιο χρειάστηκε να τροποποιήσει την απόφαση για τη συμφωνία και με το Ιράκ. Και γι' αυτό πρέπει να ξαναπεράσουμε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία συγκατάθεση. Και πάλι, ο κύριο ε, Βάινερ θα τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί είναι ε, ο Έχουμε ε, δαπανίσει 200 εκατομμύρια για το Ιράκ, έχουμε μάλλον δεσμεύσει 200 εκατομμύρια για το Ιράκ μετά από τη διεθνή διάσκεψη δωρητών στο Κουβέιτ. Είμαστε άμεσα αναμεμειγμένοι όσον αφορά την βοήθεια. Πάβο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Λίντα. δεν θα επαναλάβω τα όσα περιλαμβάνει η έκθεση της ΑΦΕΤ, δηλαδή διακυβέρνηση, κατά καταπολέμηση τρομοκρατίας, πολιτικός διάλογος, μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, μετανάστευση κτλ. Το σχέδιο χρονομοδότηση αναγνωρίζει τη σημασία της εξασφάλιση της συνέχισης ε, τη ανθρωπιστική βοήθειας ε, για την σταθεροποίηση, την ε, έγκαιρη ανάκαμψη, τη συμφιλίωση και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Καλωσορίζει την απόφαση της Ένωσης 2017 να επιλέξει το Ιράκ με από τις έξι χώρε όπου θα Π.χ. Θα, υπάρξει ανθρωπιστική ανάπτυξη ε, με επιχειρησιακές αρχές, με σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών και εξασφαλίζοντας συνεργασίες για τους στόχους της, χιλιετής βιώσιμης στόχους. Είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία αυτή, να ενισχυθεί μάλιστα παρά το ότι ε, Όλα αυτά βασίζονται σε διαφορετικούς, διαφορετικές αρχές. Ο ρόλος της χρηματο, των μέσων χρηματοδότησης The humanitarian development nexus is crucial, requires further reflection. Της, ε, της ε, υλοποίησης αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να ε, εξεταστεί και η παράταση αυτού ε, συζητείται. Ή το ξέσπασμα βίας που έχει οδηγήσει σε πάνω από 3 ε, εκατομμύρια εκτοπισμένους στο Ιράκ τονίζει τη σημασία αυτών των ανθρωπιστικών ε, δράσεων. Ε, νερό, τροφή, εκπαίδευση, απασχόληση και δυνατότητα επιβίωσης γενικότερα. Το σχέδιο γνωμοδότησης στηρίζεται στο πρόσφατο στρατηγικό διάλογο με την Κομισιόν, τονίζει την έλλειψη αποτελεσμάτων που να επιτεύθηκαν μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας και καλωσορίζει νέα χρηματοδότηση στο πλαίσιο ίσως ε, του επόμενου ενδεικτικού πολιετούς προγράμματος. Επίσης, επιβεβαιώνει τους τομείς ανάπτυξης που έχουν εντοπιστεί ως τομείς προτεραιότητας για την υποστήριξη από την Ένωση, την καλή διαχείριση της, ε, την παιδεία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών. Το σχέδιο γνωμοδότησης τονίζει τη σημασία αμερόληπτης ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξικής βοήθειας από πλευρά της Ένωσης. Το Ιράκ είναι μια πολύ ε, ε, διχασμένη κοινωνία με συνεχιζόμενες εντάσεις ανάμεσα στις παραδοσιακές ε, διαφορές ανάμεσα στους Σουνίτες, τους Ιήτες και άλλες μειονότητες, καθώς και εντός αυτών των ε, χωριστών ομάδων. Γι' αυτό και η Ένωση ε, και η βοήθειά της θα πρέπει να είναι ευαίσθητη σε αυτούς τους διχασμούς, ώστε να μην, να μην τις εντείνει τους εντείνει αυτούς του διχασμούς. Τέλος, η οικονομία του Ιράκ αντιμετωπίζει μόνιμε δυσκολίε λόγω της ασφαλ... κατάστασης ασφαλείας των ενόπλων συγκρούσεων ε, και τη διαφθορά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η Ένωση να παρέχει ε, στήριξη στο Ιράκ ώστε να οικοδομήσει δυνατότητες για να διαχειριστεί τους πόρους του και να βελτιώσει τις δυνατότητες του να επιτύχει του στόχους της χιλιετίας ε, αλλά και να ε, βελτιώσει την ισότητα. Το Ιράκ πρέπει να βοηθηθεί ώστε να δικοδομήσει δυνατότητες για την ανάπτυξη και την μεγέθυνση αναγνωρίζοντας ότι οι επενδυτέ θα παίξουν ένα άλλο και μεγαλύτερο ρόλο στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ε, αυτή ήταν η εισαγωγή λοιπόν στο σχέδιο νομοδότησης. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Εσείς κύριε Βέντς. Εγώ θα μιλήσω εκπροσωπώντας κυρία Ζαμπόρσκα η οποία κολλείεται σήμερα το Ιράκ είναι από τις χώρες κλειδιά για τη διατήρηση σταθερότητας και τη ειρήνης στην ε, Εγγύη Ανατολή. Γι' αυτό η σκιώδη συγγετριά μας δέχεται τι ε, προτάσεις του Ισηγητού για τη συνεργασία που θα συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ιράκ και βέβαια στην ε, αποκατάσταση των συνδέσμων. Η πρόσφατη ε, κατανίκηση του ηλίτα δηλαδή του Ισλαμικού κράτους ανοίγει το δρόμο. Βρίσκεται σε μια φάση όπου πρέπει το Ιράκ πλέον να σταθεροποιήσει την οικονομία του. Χρειάζεται όμως η αναπτυξιακή βοήθεια για να αντιμετωπιστούν ανθρωπιστικά προβλήματα με πολλά εκατομμύρια εκτοπισμένων πολιτών που δείχνουν ότι οι προσπάθειές μας για την ρύθμιση μετά από τη σύγκρουση δεν έχουν αποδώσει ακόμα. Υπάρχουν διάφορες ε, θρησκευτικέ κοινότητες που είδαν τους πολίτες τους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους λόγω του Ισλαμικού κράτους και που είναι πρωτίστως βέβαια πολίτες του Ιράκ. Θα είναι πολύ σημαντική ωστόσο και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει να συντονιστεί καλύτερα η ε, οργανωμένη επιστροφή των προσώπων αυτών στις συστίες τους και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια και να συμβάλλουμε με ευέλτιστες πρακτικές για να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς. Η κυρία Ζαμπόρσκα θα υποβάλει προφορική τροπολογία και αναμένει με ενδιαφέρον τον διάλογο με τον εισηγητή και με τους άλλους και όλους εισηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μακάβα. Εγώ έχω μια ερώτηση να μου επιτρέψετε να την κάνω. Έχει σχέση με αυτό που είπα και στο προηγούμενο θέμα. Δεν αναφέρεται τόσο πολύ στη δική σου έκθεση Πάβο, αλλά έχει σχέση με το Ιράκ. Σχετικά δηλαδή με το follow-up, με τη συνέχεια που δίνεται στην δικαστική συνεργασία άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβεί σε σημαντικές ανθρωπιστικές βαρβαρότητες ε, σε σημεία που από, κατέχονταν από, τον, από το Ισλαμικό κράτος. Όταν μιλούμε για εταιρική σχέση, για συνεργασία με το Ιράκ, όταν ο προηγούμενος ομιλητής μίλησε προηγούμενος, αν θυμάστε, για τους πολέμους στα Βαλκάνια και το τι έγινε μετά. Τότε είχαμε βέβαια καταστήσει όρο την ε, ε, δίκη, ε, την, το να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να εμφανιστούν ενώπιον των δικαστηρίων. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο Ιράκ. Πάπο, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Κοιτάζω όμως και προς την κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε να απαντήσετε κάτι στην ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν θέλετε δεν πειράζει, θα απαντήσει ο εισηγητής. πάω Το ζήτημα αυτό καλύπτεται στο σχέδιο εκθέσεως της Επιτροπής Εξωτερικών. Εγώ έχω επικεντρωθεί σε θέματα ανθρωπιστικά και ανάπτυξης. Και εμένα με ενδιαφέρει να ακούσω απάντηση στην ερώτησή σου, αλλά δεν ξέρω κι εγώ αν υπάρχει εκπρόσωπο εδώ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να μπορεί να πει κάτι. Νομίζω ότι ίσως να μην άκουσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερώτησή μου. Όπως στο παρελθόν είχαμε το θέμα αυτό βαριών ε, περιπτώσεων καταχρήσεων, ε, καταστατήγηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι δύο νέες γυναίκες, Γεσίντι, που ήρθαν στο ίδιο το κοινοβούλιο και μπόρεσαν να καταγγείλουν το τι έγινε και μας είπαν τότε όταν μετά από τις συγκρούσεις αυτές έρχεται η ειρήνη και αναλαμβάνει τα ενία του ελέγχου ξανά η κεντρική κυβέρνηση τι γίνεται με ε, τους δράστες αυτών των βαριών εγκλημάτων ε, θα, υπάρξουν κάποιες, θα υπάρξει κάποια απόδοση ευθυνών το θέμα αυτό ήταν βεβαίως ε, στην ημερήσια διάταξη στα Βαλκάνια όταν επανήλθε η κατάσταση. Αν δεν γνωρίζετε εκπρόσωποι της Κομισιόν μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά. Ίσως να το συζητήσουμε στα πλαίσια Τη Επιτροπής Εξωτερικών και τη Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε σαν να μην έγινε τίποτε. Η Επιτροπή λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ όμως αυτοσυστηθείτε. Ρομπέρτο Στράτσι, επικεφαλής της ομάδας Εργασία του Συμβουλίου για την Εγγύης Ανατολή. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν έχω δύο ιδιότητε. Είμαι αξιωματούχο τη Επιτροπή της Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων αλλά και επικεφαλή τη ομάδα εργασία που σα εξήγησα. Δεν είμαι εξοικειωμένο με τι λεπτομέρειε των δραστηριοτήτων που ενδεχομένω να διεξαχθούν σε σχέση με αυτό γιατί δεν είναι τη απόλυτη αρμοδιότητά μου. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι από τη σκοπιά τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Ιράκ που βασίζεται στο κοινό ανακοινοθέν τη Επιτροπή προς Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα συμπεράσματα του Ιανουαρίου του 2018 του Συμβουλίου. Το θέμα που θίγεται είναι μια από τις προτεραιότητες και αναφέρθηκε και στη συζήτηση, αναφέρεται μάλλον και στη συζήτηση που κάνουμε στην ομάδα εργασίας. Ώστε πρώτον να αχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν βλέπε και το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ για τα εγκλήματα του Νταέσ, του Ισλαμικού κράτου. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι και το ζήτημα να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ε, μεταβατικής δικαιοσύνης στο Ιράκ, ώστε να αποφευθεί ένα είδος ε, ανταποδοτικής, εκδικητική δικαιοσύνης. Καταδίκες οι οποίες να μην προέρχονται από σωστές δικαστικές διαδικασίες, και οι οποίοι θα συνεχίσουν να καλλιεργούν μια πίκρα, ιδίως μεταξύ των Σούνι, ε, διονύζοντας ένα κύκλο βίας και ανταπόδοσης. Αυτή είναι μια από τις ανησυχίες που μας διαπούν και μπορούμε να ζητήσουμε από την Υπηρεσία Εξωτερικών ε, Δράσεων να έρθει να σας μιλήσει. Στον διάλογο με τις Ιρακινές Αρχές η ανάγκη στήριξη διαδικασία αυτής είναι ένα από τα στοιχεία που συνεχίζουμε να το θέτουμε διαρκώ υπόψη του. Υπήρξαν και το γνωρίζετε εκθέσεις, αναφορές μάλλον, ανταποδοτικής βίας, ιδίως στην Ινεβή, κάτι το οποίο λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη εμείς της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων και βεβαίως και στον διάλογο με τους Ιρακινούς ομολόγους μας. Και όταν εκπρόσωποι τη Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων έρχονται στην ομάδα εργασία και συζητούμε τα θέματα αυτά περισσότερο πολιτικά, οι χώρε μέλη επιθυμούν ιδιαίτερα να δώσουν συνέχεια στα θέματα αυτά. Πρόεδρος Μακάβαν, για το θέμα που είπα εγώ, ε, δεν ήταν μαχητές του Ισλαμικού κράτους. ήταν μάλιστα ο διευθυντής του τοπικού νοσοκομείου. Άνθρωποι δηλαδή που μέσα στα πλαίσια του καθεστώτος ΝΤΑΕΣ έκαναν τέτοιες βάρβαρες πράξεις. Το ερώτημα είναι τώρα πώς αντιμετωπίζονται αυτά, αλλά να μην χαθούν από τον ορίζοντά μας. Να δούμε τι μπορείτε να κάνετε. Θα τα ξαναδούμε τα πράγματα αυτά εμείς οι γυναίκες που υπήρξαν τα θύματα ζήτησαν απόδοση δικαιοσύνης και είπαν τα ονόματα των δραστών ακριβώς επειδή θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν επιστρέφουν στο Ιράκ γιατί φοβούνται, δεν αισθάνονται ασφαλείς όσο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Καλό λοιπόν, συνεχίζει η πρόεδρος Μακάβαν, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε τίποτα άλλο να προσθέσετε πάγο, όχι. Κατάθεση τροπολογιών έως τις 2 Μαΐου του μεσημέρι έχω και ένα αίτημα. Εάν λόγω του χρονισμού, μάλλον αν θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίες, μπορείτε να το κάνετε στα αγγλικά, ώστε να ψηφίσουμε στην επόμενη συνάντησή μας στις 16 Μαΐου. Όταν ρώτησα πριν, η Ντεύκο δεν ήθελε να πει τίποτε. Τώρα θέλετε. Μάλιστα κυρία Πρόεδρε, λίγα λόγια για να πούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα είναι πάντοτε μέσα στα θέματα του διαλόγου με τις Ιρακινές αρχές. Συζητούμε τις απόψεις αυτές που όπως είπατε και εσείς είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί και η επιστροφή εκατομμυρίων εκτοπισμένων στις αιστείες τους. Και βεβαίως να λογοδοτήσουν οι άνθρωποι αυτοί με τρόπο δίκαιο, μέσα στα πλαίσια ενός δίκαιου δικαστικού συστήματος. Θα συζητούμε αυτά τα πράγματα με τις Ιρακινές αρχές. Αποτελούν άλλωστε μέρος και της τακτικής συνεργασίας μας για στήριξη της Ιρακινής κυβέρνησης για να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις και στη δική τους την ε, διοίκηση. Αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι ειδικά στοχευμένα μέτρα υπέρ των θυμάτων βιοπραγιών. Εκεί βεβαίως ε, στοχεύουμε περισσότερο. Και βεβαίως συμφιλίωση, κοινωνική συνοχή και ευαίσθητα θέματα όπως η επανένταξη των μαχητών του Ισλαμικού κράτους που θα πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι θα γίνει και επιτόπου ε, κάποια συμφιλίωση που είναι εποφελία της Ιρακινής κοινωνίας μετά από όλα αυτά τα χρόνια συγκρούσεων. Πρόεδρος Μακάμα, σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι. Ευχαριστώ τώρα. Έχουμε ένα πρόβλημα με το επόμενο θέμα, το υπαριθμό 9. Θα έχουμε ομιλητέ από το ΣΕΠΣ. Και μετά έχουμε και δύο που θα, είναι, θα μιλήσουμε για τα Trust Fund. Έχουμε τώρα και μάλλον η καλύτερη λύση είναι να ε, κάνω μια διακοπή μέχρι τις 5, δηλαδή 20 λεπτών. Εσείς όμως μου δείχνετε και το ρολόι τι συμβαίνει. Θέλετε τη Σενεγάλη τώρα. Καλώς. Να αρχίσουμε με την έκθεση αντιπροσωπείας, διότι όταν έρθουν αυτοί για τα trust fund, ναι, ας αρχίσουμε, λέει η πρόεδρος. Ήθελα να είμαι βεβαία ότι οι άνθρωποι που ήταν στις αντιπροσωπείες γνωρίζουν τα σχετικά. Να αρχίσουμε τη Σενεγάλη τότε. Μπόγκταν, εσύ πήγες στη Σενεγάλη, γνωρίζω το, 11 λοιπόν, το θέμα 11 της Το 10 αναφορά από την αποστολή στη Σενεγάλη όπου εξέτασε ιδίω τα τη εφαρμογή του Αφρικανικού Trust Fund. Ευχαριστώ. Όντως ε, αυτή η αποστολή ε, προβλεπόταν να γίνει τον Φεβρουάριο του 2017, αλλά ανεβλήθη για διάφορους λόγους και τελικά έγινε το φετινό Φεβρουάριο. Έχουμε ένα-δύο συναδέλφους ως μέλη της αντιπροσωπείας μας και ε, από την αρχή στόχοι στόχη ήταν ε, να δούμε την εφαρμογή ε, του καταπιστεύματος για την Αφρική και τα project τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί με βάση το ψήφισμα του Οκτωβρίου 2016. Το καταπίστευμα το, για την Αφρική είναι ε, το μέσο που έχουμε σε και, και ο εισηγητής για την δική μας επιτροπή ήταν ο κύριος Κοράου. Σε δυόμιση μέρες ε, συναντήσαμε τον κύριο Μακούντα που ήταν εκπρόσωπος από τον του, του Υπουργείου Οικονομίας της Σενεγάλης ε, καθώς και επίσης διάφορους οργανισμούς και ΜΚΟ που εφαρμόζουν τα προγράμματα του καταπιστέματος καθώς και τους αρμόδιους για τη συλλογή στοιχείων στο Ταμπακάντα, στη Ταμπακάντα. Μετανάστες, πρόσφυγες από την περιφέρεια του Αντίρη, γυναίκες, ε, αλλά και πρέσβεις από τις ευρωπαϊκές χώρες ε, που είναι διαπιστευμένες στη Σενεγάλη, καθώς και ολόκληρο το επιτελείο του Ευρωπαϊκού Γραφείου στο Ντακάρ που μας συνόδευσαν σε διάρκεια αυτής της αποστολής. Όπως ξέρουμε η Σενεγάλη έχει μια παράδοση ως χώρα ε, από την οποία προέρχονται μετανάστες 15 εκατομμύρια Τέσσερα-πέντε όμως ε, ε, από αυτά ζουν εκτός της Σενεγάλης και τα μισά στην Ευρώπη. Διασχίζουν τη θάλασσα με την κεντρική Μεσόγειο με σημείο κίνηση στη Λιβύη. Όλο ένα και περισσότερο. Συζητήσαμε για 10.000 κόσμο που διέσχισε το 2016 την Μεσόγειο. Το συγκρίνουμε με τη Συρία όπου είχαμε 80.000 ανθρώπους από το Αφγανιστάν, 50.000 για την Ιγυρία, που είναι επίσης πολύ περισσότεροι, δεν είναι πολύ, αλλά είναι παραδοσιακές χώρες μετανάστευσης, από τις οποίες προέρχονται μετανάστες. Οι Σενεγάλη, είναι ιδιαίτερα επικοδομητική στον διάλογο περί μετανάστευσης με την Ένωση, όμως ίσως να μην έχει καταβάλει όλες τις προσπάθειες που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί το, ε, η πανεισδοχή. Ειδικά για το καταπίστευμα, αυτό ε, αφορά τη Βόρεια Αφρική, το κέρας της Αφρικής και την ε, περιοχή Σαχέλ σε αυτήν ανήκει σε μεγάλη Την κλασική αναπτυξιακή χρηματοδότηση, το EDF, ενώ εδώ έχουμε το καταπίστευμα 3,3 δις ευρώ, μεγάλη χρηματοδότηση κυρίως από την πλευρά της Ένωσης και των κρατών μελών της και κάποιων άλλων δωρητών. Το Φεβρουάριο του 2018, 146 προγράμματα έχουν εγκριθεί για ένα σύνολο 2,4 δις ευρώ. Εστιάζεται, εστιάζονται σε δύο άξονες δράσης. Ο ένας αφορά τη δημιουργία απασχόλησης και τη διαχείριση μετανάστευσης και την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της ασφάλειας. Η αποστολή μας ήθελε να εξετάσει επί τόπου πώς διαχειρίζει, ε, διαμορφώνει ε, το καταπίστευμα αυτό τα όσα ε, χρηματοδοτεί και αν λειτουργεί εύρυθμα να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί και κατά πόσο χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση οι επαφές ε, που διοργανώθηκαν με ένα μεγάλο φάσμα εκπροσώπων με στόχο να δούμε την εφαρμογή των προγραμμάτων που στόχο έχουν να αυξήσουν την επαγγελματική κατάσταση και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση ιδιαίτερα στους νέους για μια περιοχή που παραδοσιακά ε, δείχνει ε, στέλνει μάλλον μετανάστες όχι μόνο προς την Ένωση αλλά και προς τον Τακάρ που είναι πιο, το ίδιο που είναι η πιο ανεπτυγμένη πόλη της χώρας, της Σενεγάλης. Πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική ήταν η επαφή με πρώην ε, μετανάστες από την περιφέρεια Γκαοντήρη που ήρθαν στην Ταμπακούντα για να ε, έρθουν σε επαφή με την αντιπροσωπεία μας. Και εδώ είχαμε μαρτυρίες ορισμένων από αυτούς μετανάστες ότι δηλαδή ε, τι συνέβη στο δρόμο προς τη Λιβύη και πίσω, στη Λιβύη και πίσω. Δέσμευση να επανέλθουν στη χώρα και να βρουν δουλειά και κατάρτιση ώστε να επιστρέψουν στην ε, περιοχή από την οποία προέρχονται. Επίσκεψη στο κέντρο συλλογής στοιχείων για τους μετανάστες ε, στην Ταμπακούντα δημιούργησε ε, απορίες και προβληματισμό στα μέλη όσον αφορά την αποδοτικότητά του. Γιατί έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Τη νύχτα, μόλις πέσει η νύχτα, Άρα είναι πανεύκολο οι μετανάστες να μην αναφέρουν λάθρο μετανάστες ή, ή, ή λαθρέμπορους που δεν εντοπίζονται. Δεν προβλέπεται δε κανένα ιδιαίτερο πρόγραμμα για τους ανήλικους μετανάστες. Εν γέννη ήμασταν ικανοποιημένοι με την ενημέρωση πάντως που λάβαμε από τους ε, ε, και από τους επιχειρηματίες που συναντήσαμε στην Μισήρα ε, και στην Ταμπακούντα σε σχέση με την, με τη μονάδα μεταποίησης τροφίμων. Όμως δεν ήταν 100% σαφές ότι η επίσκεψη σε αυτή την επιχείρηση, την Global Business, ήταν... Ε, μάλλον κατά πόσο αυτή η επιχείρηση έπαιρνε χρήματα από το καταπίστευμα ή αν θα έπαιρνε στο μέλλον. Ήταν πάντως πολύ θετικό να δούμε πώς παράγονται αυτά οι τροφές ε, τοπικά και πώς ε, τονίζεται η επαγγελματική κατάρτιση. Ε, διαπιστώσαμε τη δέσμευση των ε, Συνεγαλέζων νέων και στα πιο, ακόμα και στα μέρη που, από όπου προέρχεται η μεγαλύτερη μετανάστευση για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις συνθήκες διαβίωσής τους μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης. Ωστόσο, δεν είχαμε αριθμητικά στοιχεία για το πώς οι νέοι συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στον Τακάρ και οι διάφορες ΜΚΟ και από την ε, πλευρά του Λουξεμβούργου μας έδωσαν σχετικές πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά στο Σενεγάλη και το πώς αυτά χρηματοδοτούνται. Ο επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας, ο Ακίμ ε, Τουκάι συμμετείχε στις επισκέψεις ε, στην Ταμπακούντα, στην Μισήρα καθώς και στην συνάντηση που είχαμε με τον υπεύθυνο τύπο του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Ήταν πολύ θετικό που είχαμε το πρέσβη μαζί μας γιατί οργάνωσε τις μετακινήσεις καθώς και το πώς θα αρθούν τα διάφορα εμπόδια στις επαφές με τις νεγαλέζικες αρχές. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και, και το επιτελείο μας που οργάνωσε τα πάντα ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά, να δούμε και τη θετική πτυχή του καταπιστεύματος για την Αφρική, αλλά και την αρνητική για την εφαρμογή όλων αυτών. Δεν βλέπω τους συναδέλφους εδώ από την αντιπροσωπεία, κρίμα, αλλά πραγματικά ήταν ενδιαφέρον γιατί μπορέσαμε έτσι να δούμε πώς εφαρμόζονται όλα αυτά. ήταν πολύ σημαντικό να δούμε πώς γίνεται η επαγγελματική κατάρτιση, πώς επιστρέφουν οι, άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι πολύ εύκολο να επιστρέψουν. Από, περνάνε από τις μεσογειακές χώρες της Ένωσης ή από τη Λιβύη, ενώ τώρα συμμετέχουν στο Business Global, συγχετίζονται με την ασφάλεια στα τρόφιμα, σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν φτιάξει ε, αυτή την τοπική κοινότητα, χίλια άνθρωποι ζουν εκεί, έχουν πρόσβαση στην παιδεία τα παιδιά τους αλλά έχει βελτιωθεί η πρόσβαση και στο κέντρο επαγγελματική κατάρτιση. όπου μπορούν δηλαδή μετά να βρουν και δουλειά ή να ανοίξουν και μια δική τους επιχείρηση που θα λάβει ε, στήριξη από τις Ενεχαλέζικες αρχές της περιφέρειας της Ταμπακούντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. οι συνάδελφοι που ήταν στην αποστολή περίμεναν να συζητηθεί αργότερα αυτό το θέμα, γι' αυτό δεν είναι ακόμα εδώ. Μπορώ να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της DEFCO και θα προτείνω να ακούσουμε και το θέμα για την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία και να τελειώσουμε νωρίτερα τη σημερινή μας συνεδρίαση. Didier Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την αποστολή και για την ε, γενικά θετική έκθεση από τους πανευρωβουλευτές που ήρθαν σε Σενεγάλη. Μπορούμε να πούμε για το καταπίστευμα στη Σενεγάλη το έχουμε χρησιμοποιήσει και εκμεταλλευτεί από όλε τι πλευρέ του. Δηλαδή για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ε, και επαγγελματική στήριξη και στους ε, γηγενείς, δηλαδή και στους μετανάστες, αλλά και για αυτούς που παλινοστούν ή ε, που βρίσκονται στη μεταναστευτική οδό. Είναι επιτυχές λοιπόν το καταπίστευμα. καταπίστευμα. από τους λόγους είναι ότι έχουμε επικαιροποιήσει ε, παλαιότερα έργα Πρόκειται δηλαδή για έργα που υπήρχαν από το παρελθόν και σε επίπεδο κρατών μελών. Εμείς τα έχουμε βελτιώσει ε, και έτσι μπορούμε να ε, έχουμε πρόσβαση και στις κατάλληλες κοινωνικές ομάδες και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ήταν και από τους ε, στόχους του καταπιστεύματος. Άλλος στόχος ήταν η βελτίωση της επιστηστικής και τροφικής ασφάλειας σε συγκεκριμένες ε, περιοχές υψηλού κινδύνου. Αυτή η στήριξη της ανθεκτικότητας ε, είναι θεμέλια της ανθρωπιστικής βοήθειας και πολύ σημαντικά στοιχεία και για αυτούς, αυτές τις κοινωνικές ομάδες που θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν, αλλά και ιδιαίτερα ευάλωτες, ε, ιδίως ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα. Τρίτον, που αναφέρει και η έκθεση της αποστολής ότι συνδέεται με την ευαισθητοποίηση ως προς τους κινδύνους της μετανάστευσης. Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά ε, στους ε, πολίτες που θα ήθελα να μεταναστεύσουν, αλλά και για να διευκολύνουμε την επιστροφή και στο πλαίσιο του OIM ε, του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση εργαζόμαστε για αυτό το θέμα. Μετά έχουμε μια σειρά έργα που έχουν να κάνουν με τα βιομετρικά στοιχεία αλλά και με τη θέση μια εθνική υπηρεσία ταυτοτήτων ε, για να, μπορούμε, να μπορεί δηλαδή η ίδια συνεργάλη να εξετάζει και τις ροές και μια ομάδα έγκαιρης ε, παρέμβαση που συνδέεται περισσότερο με την ασφάλεια και με την τρομοκρατία ή με την ε, παράνομη διακίνηση μεταναστών. Γιατί να επενθυμίσουμε, και νομίζω το είδαν οι ευρωβουλευτές, γιατί ε, συναντήθηκαν με ε, Λίβιους μετανάστες, οι μετανάστες που έρχονταν από τη Λιβύη, όλες οι μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι υπήρχε πραγματική εκμετάλλευσή τους στη Λιβύη από τα κυκλώματα και είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση και τους διακινητές. Κάποιοι μάλιστα είναι και από τη Δυτική Αφρική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε αντλήσει διδάγματα από αυτές τις αποστολές και μπορούμε να τα διοχετεύσουμε στην επόμενη συζήτησή μας για τα καταπιστεύματα. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη νέα ε, προγραμματική περίοδο. Για να δούμε κατά πόσο θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα καταπιστεύματα και με ποιον τρόπο. Πραγματικά θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτή τη δυνατότητα. Πώς θα έχουμε την ε, πλατφόρμα επικοινωνίας πλευρές Επιτροπής και πλευρές των μελών. Το θέμα είναι ότι πολλοί μετανάστες είναι ακόμα εδώ, αλλά θα επανέρχουν. Το θέμα είναι ποιος θα επιστρέψει. Αυτές είναι μαρτυρίες αυτούς τους ανθρώπους. Χαίρονται που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οι αρχές της Ενεγάλης τους έδωσαν πρόσβαση σε γη αρχικά να έχουν πρόσβαση στην τροφή, να παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους. Χαρήκαμε που ακούσαμε και αυτές τις μαρτυρίες που λένε οι ίδιοι ότι οι διακινητές δηλαδή τους τα παρουσίαζαν όλα ρόδινα στην Ευρώπη ενώ και οι ίδιοι βλέπουν ότι δεν έχουν ούτε χρήματα, ούτε πόρους, ούτε πρόσβαση, ούτε ξέρουν πού πρέπει να αποτανθούν για να επανέλθουν, να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Είναι πραγματικά πολύ δραματική εμπειρία. Γνωρίσαμε μια νέα γυναίκα από τη, με ένα μικρό παιδί που ερχόταν από τη Λιβύη. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβαινε εκεί. Αλλά και για την συλλογή δεδομένων που ανέφερε προηγουμένω, Με αυτούς που πραγματικά Ε, δεν μπορούσαν να μείνουν στην Ευρώπη, επέστρεψαν, αλλά δεν έχουμε πλέον πρόσβαση σε αυτούς για να ακούσουμε τις δικές τους μαρτυρίες. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν που βρίσκονται εδώ δεν θα τους αρέσει, θα επιστρέψουν πίσω. Και έτσι μπορεί αυτό να αποτελέσει πολύ καλό παράδειγμα. Γιατί αυτέ οι τοπικέ κοινότητε είναι από την Γουινέα Μπισάου, από γειτονικέ χώρε, όχι από τη Σενεγάλη. Έχουν φτιάξει ε, μια αιστεία για αυτού και για τι οικογένειέ του, είναι ασφαλεί, έχουν πρόσβαση στην παιδεία και έχουν και επιστηστική ασφάλεια. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό και στο μέλλον. Για αυτού που βρίσκονται εδώ παρανόμω, αλλά θα επιστρέψουν. Βεβαίω, αν η οικογένεια κάποιου βέβαια έχει δώσει όλες τις οικονομίες της για να πάει κάποιος στην Ευρώπη, ε, φίλοι να τα καταφέρει. Αλλιώς ε, θα απογοητεύσει την οικογένειά του. Γι' αυτό και πολλοί, ακόμα και να τα πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραμείνουν. Ελένη, εξετάζουμε τώρα το σημείο για τη Σενεγάλη. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Τώρα είναι η ώρα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή. Λυπάμαι που δεν ακούσα τον κύριο Βέντα ε, σε αυτά που είπε, αλλά ήμουν στην Επιτροπή Εξωτερικών όπου συζητιόταν το ζήτημα της Κύπρου και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να, να λείψω. Ε, στη Σενεγάλη οι εμπειρίες μας ήταν σημαντικές συναντήσαμε κυρίως την δραστηριότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί αυτό κάπου έχουν γεννηθεί κάποια ερωτηματικά αν όντως δουλεύουν με το σωστό τρόπο ή αν είναι απλώς ένας τρόπος εργοδότησης ε, κάποιων ανθρώπων χωρίς να φτάνουν όλα τα κονδύλια όπως πρέπει στους ε, ε, δικαιούχους, στους αποδέχτες με τρόπο που να ε, βοηθούν την ανάπτυξη και να δημιουργούνται ε, συνθήκες ε, βελτίωσης της ποιότητας της ζωής τους. Είδαμε εντυπωσιακά πράγματα όπως τις μικρές βιοτεχνίες αλλά θα μπορούσαν με ελάχιστα χρήματα και ελάχιστη προσπάθεια να γίνουν ανταγωνιστικά ακόμη και για τα ευρωπαϊκά προϊόντα εάν υπήρχε η πολιτική βούληση να γίνει η επένδυση προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπωσδήποτε φαίνεται ότι η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για να βοηθήσει ε, στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και βεβαίως το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι ε, είναι μια χώρα στην οποία το, ε, το εμπόριο ανθρώπων δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι έχει σταματήσει υπάρχει ένα, είδος, ένα ιδιότυπο είδος τράφικινγκ κυρίως στις βορειοανατολικές επαρχίες με στόχο την διοχέτευση των ανθρώπων αυτών στην, από την υποσαχάρια Αφρική στις αχτές της ε, Μεσογείου. Το νησί που βρίσκεται έξω ακριβώς από την ε, πρωτεύουσα από τον Τακάρ είναι ένας ζωντανός ε, μάρτυρας αυτού που ακόμη και σήμερα συμβαίνει στην ε, Σενεγάλη. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπαμε, σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε για τα καταπιστεύματα εν γέννη. Οπότε και αυτά που μας είπατε και στην αποστολή ε, θα τα εξετάσουμε και στη συνέχεια στην ευαίτερη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, να αφήσουμε το σημείο 11 και να ξαναπάμε συντομία στο σημείο 10. Αποστολή στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Πήγα και εγώ μαζί με τον Νόρμπερτ Νόιζερ, που να φύγει, και ο Φρανκ Αγγέρ που δεν είναι εδώ σήμερα. Μόνο τρεις ήμασταν. Προτείνω λοιπόν να το εξετάσουμε τώρα και μετά θα δούμε το σημείο για τα καταπιστεύματα. Αφού σας παρουσιάσω πρώτα αυτή τη σύντομη έκθεση για την αποστολή αυτή. Συνιστώ στους συναδέλφους να διαβάσουν την γραπτή έκθεση που θα βρείτε στους φακέλους σας, γιατί σας δίνει μια πολύ καλή σύνοψη και της ιστορίας ε, της χώρας. Αν δεν την έχετε λάβει, παρακαλώ κύριο Σαφχάουζερ να λάβει ένα αντίγραφο της έκθεσης Νόμιζα ότι είχα ζητήσει ορισμένα αντίτυπα να υπάρχουν για τους ευρωβουλευτές. Μπορεί κάποιος να δώσει τον κύριο Σαφχάουζερ ένα αντίγραφο. Πληροφορίες λοιπόν για την ιστορία της χώρας, μία από τις φτωχότερες ε, χώρες του πλανήτη. Η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι ε, παραδοσιακά και ιστορικά αυτή η χώρα ε, ήταν υπανάπτυκτη και έπεσε θύμα και εκμετάλλευσης και αμέλειας. Υπάρχουν, υπάρχουν ορισμένες προσπάθειες να επανέλθει η ειρήνη σε αυτή τη χώρα. Η διεθνής κοινότητα έχει επενδύσει ιδιαίτερος στην χώρα αυτή όμως ακόμα υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες. Έχετε λάβει εγγραφό και του προγράμματος. Θα δείτε ότι είχαμε συνεδριάσει στο υψηλότερο το επίπεδο. Συναντηθήκαμε και με τον ε, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, ε, την Βουλή, βουλευτές, ομάδες νέων και φορείς νέων, ανθρωπιστικές οργανώσεις, Είχαμε λοιπόν την εντύπωση ότι καταβάλλονται σκληρές προσπάθειες, όμως με κάποιον τρόπο η χώρα δεν είναι ε, σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως ε, τις δυνατότητες που της προσφέρονται και στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ίσως ε, είναι καλό να διαβάσετε λοιπόν αυτή την έκθεση. Βέβαια, το πρώτο καταπίστευμα που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη ήταν ακριβώς για την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το καταστήμα Μπέκου. Πολύ γνωστό και στη χώρα αυτή. Όλοι το ήξεραν και στους δρόμους ακόμα. Γιατί βγήκαμε και στον δρόμο και συναντήσαμε ανθρώπους στην πρωτεύουσα. Μόνο εκεί μπορούσαμε να πάμε λόγω της κατάστασης ασφάλεια στη χώρα. Είναι πολύ δύσκολο να φύγει κανεί από την πρωτεύουσα. Όμως ε, στη πρωτεύουσα συναντήσαμε ε, ενώσεις γυναικών, εκτοπισμένους πολίτες που είχαν επιστρέψει στις κοινότητές τους μετά από αποτρόπαια συμβάντα πριν από μερικά χρόνια. Όλοι ήξεραν το καταπίστευμα Μπέκου και παρότι το Ταμείο Μπέκου είναι σχετικά μικρό, ε, κάπως θεωρούσαν οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ως κονδύλια υπό τον Μπέκου και το συνολικό μήνυμα ήταν παρακαλούμε βοηθήστε τη στήριξη γιατί χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Συναντήσαμε και πολιτικούς, είπα, τον πρόεδρο. που χαίρει τη στήριξη ε, του κοινού, του, του, των ψηφοφόρων, έχει εκλεγεί δημοκρατικά Είδαμε ένα κοινοβούλιο που φαινομενικά ήθελε τουλάχιστον να ε, προχωρήσει ο διάλογο, αλλά υπήρξε έλλειψη διαλόγου μεταξύ Προέδρου και ε, Κοινοβουλίου. Και οι βουλευτές ήθελαν ε, να συνεργαστούν και με ευρωβουλευτέ για να δουν ακριβώς πώς μπορούν να λειτουργήσουν ως κοινοβούλιο και πώς να αυξηθεί και η λογοδοσία του Προέδρου. Αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον για φορείς ανάπτυξης ε, και ανθρωπιστικής βοήθειας είναι πολύ δύσκολο το θέμα της ασφάλειας, είναι δύσκολο να φύγει κανείς στην πρωτεύουσα και ένα από τα βασικά αιτήματα ήταν να καταβληθούν μεγαλύτερε προσπάθειες ε, για να αυξηθεί η αίσθηση της ασφάλειας στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην χρηματοδότηση ε, και την κατάρτιση των δυνάμεων ασφαλείας με μια σειρά άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επισκεφθήκαμε λοιπόν την αποστολή αυτή και είδαμε την κατάρτιση των στρατιωτών, πραγματικά εντυπωσιακό. Είδαμε όμως και τους περιορισμούς ε, της στήριξης μας για την ασφάλεια. Α, επέθεψε ο Νόρμπερτ, ήμασταν μαζί εκεί. Είδαμε λοιπόν ότι δίνονται πολλοί πόροι στο στρατό, όμως υπήρχαν τόσοι περιορισμοί που τελικά δεν υπήρχε ούτε, ε, ούτε στολή δεν είχαν οι στρατιώτες. Κάποιοι φορούσαν πορτογαλική στρατιωτική στολή, άλλοι ιταλική, άλλοι δεν είχαν καθόλου. Δεν του έχουμε δώσει λοιπόν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ξέρω ότι αυτά είναι δύσκολα ζητήματα για την Επιτροπή μα. Αν θέλουμε όμω να εκπαιδεύσουμε ένα στρατό για να είναι σε θέση να ε, καταπολεμά ε, συμμορίε ενόπλων σε όλη τη χώρα, πρέπει να είναι ενόπλος και στρατός. Οι Ρώσοι λοιπόν τώρα έχουν λάβει εντολή από τον ΟΗΕ και εκείνοι παρέχουν τον οπλισμό στις ένοπλες δυνάμεις. Ε, υπάρχει μια ανησυχία, ένας προβληματισμός για αυτό το ζήτημα και στη χώρα και αλλού. Ο Φρανκ Έγγελ σίγουρα θα θέλει να πει περισσότερα από αυτού αν ήταν εδώ. Στο μέλλον λοιπόν θα πρέπει να δούμε καθώς ε, γίνεται λόγος και για ένα νέο ε, μέσο ασφαλείας, ότι πρέπει τα προγράμματα να βγάζουν και νόημα. Όταν καταρτίζουμε και εκπαιδεύουμε ένα στρατό, θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα χρηματοδότηση του στρατού για να λειτουργεί σωστά. Υπάρχει διεθνή κινητοποίηση και επένδυση στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Είναι πολύ δύσκολο ε, πλαίσιο δραστηριοποίηση. Πραγματικά θαυμάζω ιδιαίτερως ε, την αποστολή, τον ε, πρέσβη, το προσωπικό της ΔΕΦΚΟ, γιατί ξέρετε ότι δεν μπορούν να φέρουν συγγενείς μαζί τους, ούτε κανένας να τους επισκεφθεί. Είναι πολύ ε, αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πάλι λοιπόν εκεί. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα για να τους ε, στηρίξουμε, να τους δίνουμε μεγαλύτερα, περισσότερες διακοπές και διαλύματα και στήριξη. Έχουμε καταλήξει σε ορισμένα βήματα από εδώ και πέρα, περισσότερη στήριξη προς το Κοινοβούλιο, τη Γενική Εθνική Εθνοσυνέλευση, κάποιοι ήθελαν να επιστρέψουν στη χώρα τους για να κάνουν βήματα προς τη δημοκρατία. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεύτερον, εντολή για την ε, αποστολή ε, κατάρτισης θα ανανεωθεί φέτος. Καλό θα ήταν να κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Ευρωπαϊκή ΣΕΝΤΕ για να το εξετάσουμε και πρακτικά ζητήματα όπως προείπα. Και πρέπει να πω ότι οι συνθήκες διαβίωσης ε, των υπαλλήλων που στέλνουμε εκεί πραγματικά ήταν πολύ κακές. Εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο για να πηγαίνει και να κάνει αυτές τις αποστολές, αλλά για να το κάνουν αυτό πρέπει να τους φροντίζουμε κιόλας. Ίσως και στρεφόμενοι και προς συναδέλφους που ε, ασχολούνται και με τις χώρες ΑΚΕ και την ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης, ίσως θα μπορούσατε να τα εξετάσετε και εκεί, γιατί μία από τις, ε, ένα από τα παράπονα ήταν ο ρόλος των γειτονικών χωρών και ότι πρέπει να εξευρεθεί μία περιφερειακή λύση σε αυτή τη σύγκρουση. Καλό θα ήταν να το αναφέρετε και αυτό. Άλλο αίτημα που ακούσαμε ιδιαίτερως. Ε, ορατά σημάδια στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Θα συναντηθούμε σύντομα και με τη Φεντερίκα Μογκερίνη. Ήταν έρθει Φεβρουάριο, αλλά ήταν άρρωστη και δεν συναντηθήκαμε τελικά. Αλλά αυτό μας είπαν ότι θέλουν στήριξη από τη Φεντερίκα Μογκερίνη ή από τους επιτρόπους για να μην υπάρχει μία κόποση ε, του δωρητή. Γιατί υπάρχει αίσθηση ότι έχουμε δώσει πολλά χρήματα, έχουμε επενδύσει τόσο πολύ, αλλά και πάλι δεν βλέπουμε την πρόοδο που θα επιθυμούσαμε. Θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που διοργάνωσαν την επίσκεψη, γιατί ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διοργανωθεί και η αντιπροσωπεία εργάζεται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο κ. Σαφχάουζερ είναι εδώ, ξέρει πολλά για την χώρα αυτή. Σίγουρα θα έχει κάτι να προσθέσει. Και ο Νόρμπερτ ενδεχομένω. σα ευχαριστώ όμως ε, που διοργανώσατε αυτή την αποστολή. Ο κύριο ε, Σαφχάουζερ. Merci, Madame la, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως, πέρασα σε αυτή τη χώρα τέσσερις αποστολής πρόσφατα από το Δεκέμβριο και στο σύνολο δηλαδή έμεινα εκεί καμιά δεκαπενταριά μέρες. Ε, ήθελα να δω πάση θυσία τι μπορούμε να κάνουμε σε μια χώρα όπου σωρεύονται όλες οι δυσκολίες, διότι περί αυτού πρόκειται. Και θα αναφέρω τρία σημεία. Ασφάλεια και ανάπτυξη, ΕΚΟ και περιφερειακή ε, δυναμική. Όσον αφορά την ανάπτυξη, ε, Κάναμε μια επιχείρηση γεμάτη καλή θέληση, το λέω γνωρίζοντας τους στρατιωτικούς που ασχολήθηκαν με αυτή την κατάσταση, αλλά δυστυχώς ε, χωρίς όπλα, χωρίς στρατόπεδο. Δεν υπάρχει στρατόπεδο. οι στρατιωτικοί που εμείς έχουμε εκπαιδεύσει παλιά, παρά την καλή θέληση δεν μπορούν να είναι αποδιωτικοί. Πρέπει οπωσδήποτε δηλαδή να αναθεωρήσουμε τα μέσα. Δεν μπορούμε από τη μια πλευρά να ε, βάζουμε την ανάπτυξη και από την άλλη χωριστά την ασφάλεια και τους ε, στρατιωτικούς. Πρέπει μαζί να πηγαίνουν αυτά. Να θυμίσω ότι Αυτά που δαπανά ο ΙΕ είναι ένα δις. Για πολύ μειωμένη απόδοση, γιατί ακόμα και στον Πανγκή υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, ολόκληρα γειτονιές, τις οποίες ελέγχουν οι Σελεκά θα αρκούσε να βάλουμε μία ταξιαρχία, κινητή ταξιαρχία, που εμείς προτείναμε τρεις. Αυτή είναι μια μελέτη που κάναμε τότε με τους Ρώσους, τους Αμερικανούς και έναν ε, Γάλλο στρατηγό. Να βάλουμε δηλαδή ένα, ένα κινητό τάγμα ε, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Το κόστος αυτού του τάγματος πέρα από τα όπλα ήταν 60 εκατομμύρια, ε, ε, εκατομμύρια ευρώ και ετήσιο κόστος με τη βοήθεια των καλύτερων ειδικών ήταν γύρω στα 20 εκατομμύρια. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι δαπανάν, δαπανά ο ΙΕ και τι θα μπορούσαν να κάνουν τρεις δυνάμεις που έχουν αναλύσει την κατάσταση. Γαλλία, δηλαδή Ρωσία και ΙΠΑ και που λένε ότι με ένα τάγμα κινητό με 850 ανθρώπους Εκεί κανονικά θα έπρεπε για ολόκληρη τη χώρα να υπάρχουν τρία-τέσσερα τάγματα τέτοια κινητά θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε απολύτω την ασφάλεια. Απολύτως πρόκειται για επαγγελματίες στρατιωτικού, γνωρίζουν για την πράγμα μιλάμε, που έχουν τη συνήθεια της δράσης και ε, το λένε αυτό. Πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε γιατί δεν τα καταφέρνουμε, γιατί έχουμε μπλέξει σε διαδικασίες που δεν το επιτρέπουν. διότι αυτό που κάνει ο ΙΕ δεν είναι αποτελεσματικό, ούτε στην Κεντρική Αφρική, ούτε είναι στο Κονγκό, ούτε στο Μαλί. Γιατί ε, αποτυχάνουμε λοιπόν και γιατί δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ενώ όταν έχουμε τις τρεις δυνάμεις που μπορούν να παρέμουν, οι στρατιωτικοί σας λένε πολύ καλά τι πρέπει να γίνει και ποιο είναι και το κόστος. Το καταπίστευμα Μπέκου. Ήσασταν εκεί δύο μέρες εγώ 15. Ακούστε. το ελεγκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και οι παρατηρήσεις του είναι κέρυες. Λένε τι, ότι το κράτος θα πρέπει να συνεργαστεί, που δεν συνεργάζεται. Ακόμα και σας λένε το αντίθετο. Έχω έρθει σε επαφή με τους επικεφαλείς, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Συντονισμού, τον Υπουργό Αμήνης. 15 ώρες περίπου ε, συνομίλησα με τον Υπουργό Αμήνης. Το καταπίστευμα Μπεκού δεν είναι σωστό, δεν είναι προσαρμοσμένο. Βοηθά τις ΜΚΟ και τις αναπτυξιακές, ε, τους οργανισμούς. Δεν συνεργάζεται με το κράτος. Όμως δεν μπορείτε να κάνετε και το λέω και το ξαναματαλέω. Δεν μπορείτε να κάνετε ανάπτυξη χωρί τη στήριξη την κυβερνητική. Η κυβέρνηση είναι έξω από το κύκλωμα του καταπιστεύματο Μπέκου και όταν προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπεύθυνη να προσαρμάσει αυτό το Μπέκου λέει πως δεν γίνεται. Ο κύριος Μανσερβισή μου έλεγε πως γίνεται και έχω κάνει νέο ραντεβού μαζί του. Η υπεύθυνη μου λέει πως δεν γίνεται. Εάν δεν είναι δυνατόν, εγώ που είχα κινητοποιήσει 100 εκατομμύρια από ιδιωτικά χρήματα για να συνοδεύσουν τα δημόσια χρήματα, δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Δεν πάω άλλο εκεί γιατί για την ώρα το σύστημα έχει μπλοκαριστεί. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό, με ιδιωτικά χρήματα το τμήμα το, δημόσιο, το ιδιωτικό και το ε, δημόσιο επιπλέον. Πρέπει επίσης εκ των προτέρων να ρυθμίσουμε γιατί οι επιχειρήσεις που θέλαν να έρθουν με εγκατέλειψαν λόγω ασφάλειας. Εφόσον δεν υπάρχει ασφάλεια στον μπανκί, δεν γίνεται να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Δεύτερον, όμως διαρθωτικά θα πρέπει το καταπίστημα βαϊκού να δουλέψει όχι μόνο να συνεργαστεί με το κράτος, να είναι ένα καταπίστημα όπου το κράτος της Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας να συμμετέχει στη διαχείριση και στην οργάνωση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε κάθε ευθύνη για να πει ότι είναι έτοιμος να, συντάξει, να συστήσει μια ad hoc επιτροπή όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι για την ανάπτυξη σε αυτή την ad hoc επιτροπή ώστε όλα αυτά να γίνουν με πλήρη διαφάνεια. Δυστυχώς η επιτροπή μας είπε πως αυτό δεν γίνεται. Αντίθετα με τον ε, Διευθυντή Υπεύθυνο για την Ανάπτυξη που είναι πολύ πιο ευέλικτος και που είναι και πίσω από την Κομισιόν. Πρέπει να αποφασίσουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τώρα, Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί όσον αφορά την ασφάλεια αν δεν υπάρχει περιφερειακή δυναμική. Τι κάνουμε, ποια βοήθεια δίνουμε για να υπάρξει τέτοιου είδου δυναμική. Βεβαίως έχουμε το G5. Αλλά η ε, Κεντρική Αφρική δεν είναι μέλος τι κάνουμε με το Καμερούν, τι κάνουμε με το Κονγκό, τι, πώς έχουμε μια, μια γενική προσέγγιση για την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Δεν θα έπρεπε να δοθούν πιστώσεις ώστε πραγματικά να στηθούν projects για μια τέτοια περιφερειακή δυναμική. Αυτό είναι το θέμα που είχαμε την περασμένη φορά. Βλέπουμε πώς λειτουργεί αρκετά καλά προς την ακτή του Ελεφαντοστού και τη Δυτική Αφρική, ενώ στην Κεντρική Αφρική δεν υπάρχει τέτοιου είδου ε, περιφερειακή δυναμική. Έχω έρθει σε επαφή με το παλαιότερο ηθήνοντα τώρα μου διαφεύγει το όνομά του και μου έλεγε ότι ε, δεν λειτουργεί το πράγμα ακριβώ επειδή δεν υπάρχει και περιφερειακά δυναμική. Εγώ είμαι απεσιόδοξο, ε, κυρία Πρόεδρε. Είμαι απεσιόδοξο γιατί τα πράγματα γίνονται όπω το είχα προβλέψει. Έλεγα το Δεκέμβριο πω η κατάσταση σε θέματα ασφάλεια θα επιδεινωθεί και επιδεινώνεται. Έλεγα πω δεν έχουμε μέσα κατάλληλα και αυτά τα μέσα δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα και αν ο Διευθυντής της Ανάπτυξης εδώ ακριβώς μου είπε και έχω το βίντεο που κυκλοφόρησε να φτιάξουμε τα διευθυντικά ταμεία σε εταιρική σχέση μαζί με την κυβέρνηση αν είναι αυτό απαραίτητο. Η εφαρμογή δεν γίνεται και αν δεν εφαρμοστούν όλα αυτά αυτό σημαίνει πως όλα τα project που εγώ προετοίμασα με την κυβέρνηση το δημόσιο τμήμα των όσων μπορούν να φτιαχτούν και να οδηγήσουν και σε ιδιωτικέ επενδύσεις δεν θα δούνε το φως της ημέρας και οι ιδιωτικέ επενδύσεις δεν πρόκειται να αναλάβουν όλο αυτό το, το κομμάτι των επενδύσεων, να πρόκειται για την ηλεκτροδότηση ή για σφαγεία ή για δρόμους, όλα τα πάντα. Πώς όλα αυτά θα αποδώσουν και επιπλέον δεν υπάρχει και ασφάλεια. Και τρίτον, και επανέρχομαι, δεν υπάρχει περιφερειακή δυναμική που είναι θεμελιώδης για την ασφάλεια βεβαίως. Και ήμουν με τον εκπρόσωπο της ασφάλειας του Καμερούν έκανα μία αποστολή γιατί τον γνωρίζω πολύ καλά αυτή τη χώρα ε, πριν από 10-15 χρόνια εκεί ε, παρενέβη πολύ αλλά δεν υπάρχει όπως σας λέω περιφερειακή δυναμική για την ασφάλεια άρα δεν υπάρχει και ασφάλεια. ανάπτυξη του Μπαγκή σταματά στα σύνορα. Πώς θέλετε να σκεφτείτε την ανάπτυξη του Μπαγκή χωρίς να αναπτυχθεί ολόκληρη η ζώνη 400-500 σε ακτίνα 400-500 χιλιόμετρων όπου είσαι αμέσω βρίσκεστε σε άλλες χώρες. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά πραγματικά εγώ βάζω την καρδιά μου σε αυτή την υπόθεση και εκφράζω εδώ την απελπισία μου, σας το λέω. Ελπίζω πως παρόλα αυτά θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος Μακάβαν θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει βέβαια το Μπέκου Φαντ, αλλά και είπε το CDF Fund. Αν τα νούμερα του EDF είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερο και είναι για την στήριξη των δημοσίων υπηρεσιών. Έχουμε αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Δεν είμαι βέβαια λοιπόν ότι θα έχουμε παρόντες, του εκπροσώπου της Επιτροπής στην κατάλληλη στιγμή. Α, ε, ο συνάδελφό μα θέλει να λάβει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ορισμένα πράγματα τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή μου. Ποτέ δεν έχω βρεθεί σε χώρα όπου οι καταστροφές στην πρωτεύουσα από τον εμφύλιο πόλεμο και από τις αναταραχές να είναι τόσο ορατές και εκτεταμένες. Υπάρχει ανάγκη βελτιώσεων Έχουμε και τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τα Ηνωμένα Έθνη που με την ε, προσπάθειά τους έχουν βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό που βλέπω να λείπει είναι το στοιχείο της ασφάλειας. Ο κ. Σαφχάουζερ επίσης το ξεκαθάρισε αυτό στην παρέμβασή του. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ανάπτυξη. Ασφάλεια είναι εγγυημένη μόνο σε τμήματα της πρωτεύουσα. Τώρα, πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, ποιον ρόλο θα πρέπει να παίξουν τα Ηνωμένα Έθνη και μάλιστα ενισχυμένα, ποιες ε, ενδεχομένως ε, εντολές θα πρέπει να δοθούν από τα Ηνωμένα Έθνη προς την ε, Γαλλία ή προς άλλες χώρες μέλη οι οποίες δείχνουν ιδιαίτερη δέσμευση εκεί. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Για το budget support, για την δημοσιονομική στήριξη που ρωτήσαμε μας είπαν καθαρά ότι χωρίς δημοσιονομική στήριξη δεν θα υπάρχει καν κράτος. Ε, ολόκληρο το οικοδόμημα είναι τόσο εύθραυστο που το χρειάζεται αυτό απολύτως για να μπορέσουν να διατηρήσουν κάπως τις κρατικές δομές ώστε να έχουν κυβέρνηση και ε, ε, κοινοβουλευτικό σώμα. Για την training mission ο κύριος Βέντα είπε τα πιο σημαντικά και εδώ ήταν τρομακτικό που είδαμε πόσο ενθουσιώδεις είναι οι εκπαιδευτές που έχουμε αποστείλει εμείς οι ίδιοι εκεί, αλλά πόσο δύσκολες και σκληρές είναι οι συνθήκες διαβίωσης. Είναι απίστευτο που οι άνθρωποι αυτοί αντέχουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτή την training mission και εξ αντιστρόφου και οι εκπαιδευόμενοι είναι και αυτοί οι ενθουσιώδεις αλλά τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Είδαμε ασκήσεις είδαμε ασκήσεις ε, τακτικών κινήσεων χωρίς πυρομαχικά. Πιο πολύ φαινόταν σαν ε, παιχνίδι παιδιών που παίζουν με ξύλινα όπλα. Ε, εμένα με πόνεσε η καρδιά μου. Χρειάζεται να τους διατεθούν τα αναγκαία μέσα. Ε, ε, επίσης ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν για μας το γεγονός ότι η Ρωσία η οποία σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική ήταν λίγο, ήταν περιορισμένα παρούσα, ξαφνικά βρίσκεται τώρα εκεί και εξοπλίζει τον στρατό ή τέλο πάντων δηλώνει την πρόθεση να εξοπλίσει τον στρατό. Εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπατε κύριε Σαφχάουζερ, αλλά δεν κατάλαβα καλά με ποιον ρόλο με ποιον ρόλο ε, βρίσκεστε εσείς επιτόπου στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ως ιδιώτης σας έχουν αποστείλει επιχειρήσεις, συνεργάζεστε εκεί με επιχειρήσεις. Ε, δραστηριοποιήστε κατ' εντολή της γαλλικής κυβερνήσεως. Όλα αυτά για μένα είναι ασαφή, πολύ ασαφή. Έστω και αν ε, βρίσκω ότι ίσως έχετε δίκιο σε ορισμένα οσιώδη πράγματα, όταν λέτε εμείς ή όταν λέτε εγώ, ε, ποιοι, ποιοι είστε αυτοί και από πού ε, λαμβάνεται αυτή την... Ε, πώ αναλαμβάνει αυτή τη δράση ο κύριος Σαφχάουζερ. Κοιτάξτε, 20 χρόνια ήμουν επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνεργασίας, το οποίο δραστηριοποιείται στη ζώνη αυτή. Δεύτερο, πράγματι έχω εκτελέσει, έχω εκτελέσει αποστολές της γαλλικής κυβερνήσεως. Τρίτο, ήμουν στο πρόγραμμα ε, για την Αφρική της Παγκόσμιας Τράπεζας. Επομένως είχα εκεί αποστολή μαζί με Γάλλους εκπροσώπους οι οποίοι δουλεύουν για την ε, ε, ασφάλεια σε συνεργασία με στρατιωτικούς. Το λέω καθαρά. Δεύτερο, ως ιδιώτης και επειδή είμαι πεπισμένος ότι χρειάζεται να εμφυσιθεί μια δυναμική ε, τα ταμεία επενδύσεων για να προωθηθούν οι ιδιωτικές επενδύσει, προσπάθησα να κινητοποιήσω ανθρώπους που δραστηριοποιούνται ε, στις επενδύσει, προσπάθησα να το κάνω στη συνεργασία με μια ε, εταιρεία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Εμμυράτα και όπου συγκεντρώνει ε, διαφόρους και από την Ευρώπη και από τη Γαλλία, αλλά όχι μόνο από τη Γαλλία, αλλά και ανθρώπους από τα Ενωμένα Εμμυράτα και προσώπους των Ηνωμένων Εθνών και ανθρώπους που έρχονται από την Ασία για να δούμε με όλους αυτούς μαζί τι μπορούμε να κάνουμε για να φτιάξουμε ένα ε, ταμείο επενδύσεων ιδιωτικό. Αυτά τα εξήγησα και στον Διευθυντή Αναπτύξεως. Έκανα μία έκθεση όλων αυτών των προσπαθειών μου. Αυτό που χρειάζεται από την άλλη μεριά ως δημόσια επένδυση. Χρειάζεται και στήριξη των δημοσίων επενδύσεων. Βεβαίως για να λειτουργήσουν και ιδιωτικέ επενδύσει. Το πιο σημαντικό το είπατε, είναι η ασφάλεια. Γύρω από κάποιο project ασφαλώ πρόκειται πρωτίστω για δημόσιε επενδύσει. Αλλά οι δημόσιε επενδύσει είναι αναγκαίε και για να υπάρξουν και ιδιωτικέ επενδύσει. Εγώ σα τα είπα αυτά προηγουμένω και ανατομέα ξεχωριστά. Προηγουμένω ήμασταν μόνο ο κ. Βέντα και εγώ εδώ παγόντες Τώρα όμως ε, έχουμε πολύ περισσότερους ενδιαφερομένους ευρωβουλευτές και επομένω παίρνει περισσότερο χρόνο. Μου είπαν ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Επιτροπής είναι παρούσα και θα ήθελε να απαντήσει. Μάρτιν Κάουντα από την DG DEFCO, Development Cooperation δηλαδή, και μετά να προχωρήσουμε για την, ε, με την μελέτη για τα Trust Fund. Όπως είπα, έχουμε ανατρέψει λίγο το πρόγραμμα της ε, ημερήσιας διάταξης σήμερα. Ορίστε λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την αποστολή που εκτελέσατε εκεί και την επίσκεψή σας και τη στράτευση που δείχνετε για την κεντροαφρικανική ε, υπόθεση που είναι πάρα πολύ σημαντική για ολόκληρη την αντιπροσωπεία μας. Ε, χαιρόμαστε πολύ για τις ε, εκθέσεις που έχετε συντάξει που δείχνουν πραγματικά ποια είναι η εικόνα και η, πραγματικά, και και συνεχιζόμενη ε, δέσμευση εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε και για τα σχόλια που κάνατε για τους τρόπους, για τους όρους διαβίωσης των ε, εκπροσώπων μας εκεί. Τα οποία σχόλια θα τα μεταφέρουμε στα πρόσωπα που ενδιαφέρονται. Ήθελα λοιπόν να είμαι πάρα πολύ σύντομη, περιορίζομαι σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, τη ΕΚΟ. Άλλος κανείς. Υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα ε, σημεία follow-up, τα οποία θα θέσουμε και υπόψη της κυρίας Μογκερίνη. Αν μπορέσουμε θα οργανώσουμε συνάντηση μαζί της για να θέσουμε υπόψη τα θέματα αυτά, γιατί βεβαίως το νόημα των αποστολών αυτών είναι να διδαχθούμε από αυτές αλλά και να θέσουμε ε, τα θέματα και να μπορέσει να υπάρξει και κάποιο κάποιος μηχανισμός χρηματοδότησης των ζητημάτων ασφαλείας και κυρίως ε, στολές για στρατιώτες και εξοπλισμός. Ε, να αφήσουμε τώρα το υπαριθμό 10 και να επανέλθουμε στο 9 νομίζω έτσι είναι. 9 για τη Σενεγάλη και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία τα οποία συνδυάζονται με τούτο εδώ. Το 9 δηλαδή εποπτεία των Trust Fund Παρακαλώ τους επισκέπτες να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Έχουμε μελέτα, μελέτη συγγνώμη, από το ΣΕΠΣ για την δημοκρατική λογοδοσία, πρακτικές και ε, προκλήσεις για τα Trust Fund που έχει ήδη, έχουν ήδη υποβληθεί στις ε, άλλες συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Έχει ενδιαφέρον η έκθεση και νομίζω ότι θα είναι και χρήσιμο για τους ε, συναδέλφους να ακούσουν ορισμένα από τα θέματα αυτά τα οποία συζητήθηκαν στη συνάντηση αυτή της Επιτροπής Προϋπολογισμών όπου μου φάνηκε ότι δεν έδεσαν αρκετό χρόνο στους ε, ε, ομιλητές διότι οι βουλευτές είχαν δεσμεύσει από 10 λεπτά για τον εαυτό τους Γι' αυτό εγώ δεν θα μιλήσω περισσότερο. Έχει, έχει διανεμηθεί η μελέτη την οποία θα παρουσιάσουν. Έχετε δώσει αντίγραφα στους συναδέλφους μου. Υπάρχει μόνο μία online version. Μπορείτε να το στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στείλτε το στους βουλευτές. Έχουν όλοι τα iPad τους ή τους υπολογιστές τους μαζί για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να ζητήσουμε από τους προσκεκλημένους μας, η κυρία Βοσιλούτε πρώτη και ο κύριος Νούνιες, θα παρουσιάσουν τα πιο σημαντικά συμπεράσματα. Όταν τους άκουσα πρώτη φορά εγώ στην άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή, μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα αυτά. Ε, για το αν υπάρχουν trust fund, θα πρέπει να υπάρχουν όπως το Beku Fund, για ιδιαίτερες συνθήκες ή θα χρειαστούν περισσότερα όπως το Africa Trust Fund ή αν θα πρέπει να ε, συγχωνευτούν στο mainstream. Ποιος από τους δυο θα ήθελε λοιπόν να αρχίσει εξ ημών. Ε, thank you, Madam. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές που είναι εδώ και τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημιουργήσαμε αυτή τη μελέτη για τα ευρωπαϊκά καταπιστεύματα και επικεντρωθήκαμε κυρίως στην εποπτεία, τη διαχείριση καθώς και την θέσπιση των καταπιστευμάτων. Okay. Does it work? How it works? Sorry? How it works? Oh, I don't know. Somebody, Carol, can help? help? Okay, good. Ah, okay, good. Ah, okay, okay. Okay. Um, yeah, so the scope... Το πέντε εφαρμογή της μελέτης αφορούσε τα στοιχεία που βλέπετε. από την ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Εκεί λοιπόν έχει παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, καθώς ε, και στην Επιτροπή Προπολογισμών του Κοινοβουλίου. Είναι η τρίτη φορά λοιπόν που την παρουσιάζουμε. Χαιρόμαστε που υπάρχει τόσο ε, έντονο ενδιαφέρον για την μελέτη μας. Αποτελεί αντικείμενο συλλογικής προσπάθειας. Δύο, δύο μονάδες ε, του ΣΕΠΣ έχουν ε, ενεργήσει από κοινού για αυτή τη μελέτη. Βλέπετε εδώ και τους συντάκτες. Ο Χόρχε θα πάρει το λόγο στη συνέχεια για να σας παρουσιάσει την εμπειρία από άλλα καταπιστέυματα φορέων όπως ο ΙΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Κατά τη δική μας ε, εκτίμηση της διακυβέρνησης και της εποπτείας, επικεντρωθήκαμε σε τέσσερα καταπιστεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα έχουν ε, κατονομαστεί ως ε, επίγουσας ε, βοήθειας ή βοήθειας μετά από μια κρίση. Και υπάρχει και ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, ε, η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, ο σχετικός μηχανισμός. Θεωρήσαμε ενδιαφέρον να τα συγκρίνουμε και να εξετάσουμε τυχόν κοινά ε, στοιχεία μεταξύ των καταπιστευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μέσου για τους πρόσφυγες στην Τουρκία που εντάσσεται στο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε γιατί υπήρξε πολιτική προτεραιότητα μετά την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θέλουμε να δούμε την προσταθμένη αξία και μετά από την ε, υιοθέτηση της πολιτικής του ευνομοθετήν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιωθεί και ως δημοσιονομική αρχή και ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε η πορεία των καταπιστευμάτων εδώ. Κάποιες φορές βέβαια είναι δύσκολο να δούμε την κατάσταση επιτόπου. Θέλαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι δεν ήταν ένας ε, λογιστικός έλεγχος, αξιολόγηση αντικτύπου ή ποιοτική αξιολόγηση των έργων. Όμως λάβαμε υπόψη ιδίως ε, την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί βρήκαμε σημαντικά στοιχεία εκεί. Τι μεθόδους ε, χρησιμοποιήσαμε. Ναι, μπορούν αυτά να τα διαβάσουν οι συνάδελφοι αν θέλουν. Okay. Okay, we want... Παρακαλούμε να περάσετε στην ουσία της μελέτης. Ναι, αλλά θέλαμε απλώς να τονίσουμε ότι ήταν μια διαδραστική διαδικασία. και ότι καλύψαμε εξελίξεις μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει τώρα νέες αιτήσει εκθέσεις, ωστόσο τότε δεν τις είχαμε όταν κάναμε τη μελέτη δεν σταθήκαμε μόνο στα διαθέσιμα στοιχεία που μπορούσαμε να βρούμε και στο διαδίκτυο και σε επίσημα έγγραφα, αλλά είχαμε και συζήτηση της ομάδας ε, με την κοινωνία των πολιτών και οργανώσεων που ε, εποφελούνται των καταπιστευμάτων για να δούμε τι συμβαίνει στην πράξη Λοιπόν, ε, στην παρουσίαση θα σταθούμε περισσότερο στο καταπίστευμα για την Αφρική που συνδέεται στενά με την ε, Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής στη Βαλέτα. που βασίζεται βέβαια σε περιπτώσεις έκτατης ανάγκης, οπότε είναι δύσκολο για το Κοινοβούλιο να ε, ασκήσει δημοκρατικό έλεγχο εξάντε. Και θα μείνουμε και στο καταπίστευμα Μπέκου. Επίσης είναι ένα καταπίστευμα έκτη της ανάγκης ε, που βασίζεται στο EDF. Εξετάσαμε τους όρους θέσπισης. Ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι σαφής ότι τα καταπιστεύματα δίνονται να συσταθούν είτε ε, για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είτε post-emergency, δηλαδή κατόπιν της έκτακτης ανάγκης, ως ανταπόκριση δηλαδή σε αυτές. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κλείνει ε, συμφωνίες κατόπιν εξουσιοδότησης ή να έχει και θεματικές ενέργειες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να δίνει προκαταβολικά την συνέντευξή του. Επίσης, από τον κανονισμό προκύπτει ότι θα πρέπει να ε, καταδεικνύεται η προσθεμένη αξία του καταπιστεύματος και να συνάδει με άλλες ε, αρχές όπως δημοσιονομική διαχείριση, διαφάνεια, λογικότητα και το καθεξής. το σκεπτικό και ο στόχος ε, των καταπιστευμάτων ήταν και να αυξηθεί η προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις χώρες, καθώς ε, και η πολιτική ορατότητα και προβολή των κρατών μελών Ακούσαμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και έτσι ε, είναι δυνατή η ταχύτατη υιοθέτηση αποφάσεων, όμως είδαμε στη μελέτη μας ότι όταν αυτό ισχύει για την έγκριση έργων, οι φάσεις διαπραγμάτευσης μπορούν να καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο από ότι στους ε, συνήθεις χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, όπως ε, ε, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Κάτι που είναι σημαντικό και θέλουμε να το τονίσουμε είναι ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ενεργοποιούνται εν καιρό κρίσης. Και έτσι αναφέρεται και η έκτακτη φύση τους, ας πούμε. Αυτό που επισημαίνουμε εμείς είναι τα καταπιστεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πλέον κατάλληλο μέσο σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις όταν υπάρχουν πιεστικές ανάγκες. Η σύσταση του καταπιστεύματος Βέκου είδαμε ότι το στήριξε και η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου ότι δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία επίσημη αξιολόγηση για την θέσπιση αυτού του καταπιστέυματος... ούτε υπήρχε ε, σαφής και ολοκληρωμένη ανάλυση των αναγκών. Ωστόσο, το ελεγκτικό συνέδριο θεωρούσαν ότι καλώς ε, συστάθηκε το ε, καταπίστευμα δεδομένη τη κατάστασης, γιατί η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία ε, υποχρηματοδοτεί το και τα αναπτυξιακά προγράμματα ήταν πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε στον ΟΣΑ αναφερόταν ως ορφανή από ενίσχυση. Και υπήρχε και το θέμα της μεταβατικής, της μετάβασης από τη μία κυβέρνηση στην άλλη. Και έτσι το... το ενδέκατο ενδεικτικό πρόγραμμα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν αναφέρθηκε ότι ε, κατ' εξαίρεση το καταπίστευμα Μπέκου μπορούσε να συσταθεί. Όμως, το ελεγκτικό συνέδριο και εμείς λέμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνει ε, η συνήθις διαδικασία. Αναφέρθηκε λοιπόν πολλές φορές ότι το καταπίστευμα συστήνεται ενώ υπάρχει μία πλειάδα άλλων καταπιστευμάτων και άλλων μέσων χρηματοδότησης αναπτυξιακής Οπότε για να μην ε, συγχέονται και να μην δημιουργείται σύγχυση και μπέρδεμα ε, και στους δικαιούχους και σε αυτές τις χώρες, θα πρέπει να αποφεύγουμε αυτές ε, τις λύσεις. Έτσι καλλιώς αναφέρεται ότι πρέπει πάντα ε, να τηρείται και το κριτήριο της προσθετικότητας. Ήταν δύσκολο όμως να παρακολουθήσουμε και την ε, ε, συνεχιζόμενη υλοποίηση των έργων γιατί δεν υπήρχε σημείο αναφορά benchmarking για να καταλάβουμε και εμείς ακριβώς τι χρησιμοποιούμε σημείο αναφορά για να τα αξιολογήσουμε. Τώρα, το καταπίστευμα για την Αφρική. Και αυτό δημιουργήθηκε ως ε, κατεπήγον ε, καταπίστευμα. Καλύπτει σχεδόν τη μισή Αφρικανική Ήπειρο και δημιουργείται το ζήτημα ποια ήταν η κατεπήγουσα κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το καταπίστευμα. Στην αρχή δημιουργήθηκε για την περιοχή του Σαχέλ, του Τσάντ και μετά το, για το κέρας Αφρικής και τη Βόρεια Αφρική. Αυτά προσθέθηκαν στη, στην πορεία. Αυτό είναι προφανές ακόμα και σήμερα και λέμε ότι στο Τσάντ και στο Σαχέλ Ε, δόθηκε έμφαση στην μετανάστευση και στην ανάπτυξη, όμως ε, τώρα με τη νέα εταιρική σχέση το Τσάντ και το Σαχέλ επίσης μπαίνουν ε, στο προσκήνιο. είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι ε, βασικές αιτίες ε, της μετανάστευσης είναι ουσιαστικά γενός ένα αναπτυξιακό ζήτημα και θα πρέπει να καλύπτονται και να αντιμετωπίζονται με έναν ε, αναπτυξιακό μηχανισμό, όπως είναι το EDF ή το DCI. Τα ενωσιακά καταπιστεύματα έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια. όπως αναφέρεται και στο δημοσιονομικό κανονισμό. Όμως αν θέλουμε να υπάρχει η ανάπτυξη, αυτό γίνεται με βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Δεν γίνεται να επαφείται αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια μόνο στη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Αυτό είναι κάτι που επισημάναμε στη μελέτη μας. το καταπίστευμα για την Αφρική είδαμε ότι αν σκοπός είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού, ιδίως έμφαση δίνεται ε, στο κέρας Αφρικής και στη Βόρεια Αφρική, αυτό καλύτερα θα μπορούσε να ε, ενταχθεί σε ένα θεματικό καταπίστευμα, ακόμα και ξεχωριστά. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα για τη διακυβέρνηση και τη λογοδοσία. Σημαντικό είναι να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ρόλο παρατηρητή και σε συμφωνίες και σε επιχειρησιακές επιτροπές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να ασκήσει δημοκρατικό έλεγχο και ε, προσκαλείται σε στρατηγικά συμβούλια, όμως τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου δεν χρησιμοποιούν πάντα αυτή τη δυνατότητα, δεν την αξιοποιούν. Κάποιες φορές υπάρχουν και ζητήματα πρακτικά ολομέλειας του Στρασβούργου, ενώ οι συνεδριάσεις γίνονται στις Βρυξέλλες, άλλες φορές γίνονται και αλλού ακόμα και στις ε, χώρες προορισμού αυτών των ε, ταμείων. Okay, Mm. So we found that uh, most important issues are the ongoing uh, τα πλέον σημαντικά ζητήματα σε ό,τι αφορά ε, την εξάντε και συνεχιζόμενη ε, δημοκρατική λογοδοσία. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στα προγράμματα που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν, χρηματοδοτηθούν σε επιτροπές όπου δεν εκπροσωπείται το Κοινοβούλιο και είναι μια εκτελεστική αρμοδιότητα, όμως ε, θεωρούμε σκόπιμο αυτή η διαδικασία να καταστεί πιο διαφανής. Ιδίω ό,τι αφορά, ε, ιδίω εφόσον φορείς του ΟΗΕ και άλλων καταπιστευμάτων ε, μπορούν να παρακολουθήσουν όσους παρατηρητές. Για την έξπος δημοκρατική λογοδοσία, ξέρουμε ότι υπάρχουν ετήσιες εκθέσεις και τι λογαριασμοί που υποβάλλονται προς το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και μηνιαίε και εξαμηνιαίε εκθέσεις. Το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ασκήσει δημοκρατικό έλεγχο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια τη διαδικασία απαλλαγή. Mm-hmm. Um, so we found it uh, difficult that it's. Uh, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανησυχητική τάση ε, θέσπισης και άλλων καταπιστευμάτων. Ξεκίνησε ως ε, ε κατεπίουσα διαδικασία, αλλά βλέπουμε ότι παγιώνεται, ιδίω στον τομέα τη ανάπτυξη. Ιδίω η Υπουργοί Εσωτερικών και αυτή η λειτουργία κάπως ε, υπησέρχεται μέσα στην ευρύτερη λειτουργία του συστήματος. Yes, let me just continue a moment because we, we are... Να συνεχίσω εγώ μια στιγμή αν με επιτρέπετε. Αυτά που ακούσαμε ως τώρα είναι κάποια από τα θεμελιώδη θέματα. Γιατί δημιουργήθηκαν τα trust fund. Είναι μέγα ερωτηματικό. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ένα πολλαπλασιασμό των trust fund παντού, εκτός, της, ε, εκτός του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ούτως ή άλλως η EDF λειτουργεί εκτός. Αλλά βλέπουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή χρησιμοποιούνται διαδικασίες CDF για να φτιαχτεί ένα trust fund το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει μετά και κοντή δικά της. Και βλέπουμε και ένα μηχανισμό όπως ο EDF που επιτρέπει να υπερβούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με trust fund από αλλού. Δηλαδή κάποια trust fund προκαλούν κάποιες εντάσεις και φαίνεται πως θα υπάρξουν και άλλα trust fund στο μέλλον. Τώρα προέρχεται και ο προπολογισμό. Εγώ έχω να τονίσω το εξή. Πρόκειται για κάτι που πρέπει να ελεγχθεί. Ποιο είναι ο λόγος για τα trust fund, λόγω έκτακτων καταστάσεων, λόγω του ότι υπάρχουν περισσότερα χρήματα, λόγω του ότι οι χώρες μέλη θέλουν άμεση πρόσβαση στα χρήματα αυτά. Εμείς το βλέπουμε αυτό διαμορφώνεται ως τάση. Και τα Ηνωμένα Έθνη και οι χώρες των Ηνωμένων Εθνών δηλαδή προτιμούν να χρηματοδοτούν συχνά μέσω ενό trust fund, γιατί αυτό του δίνει μια διαφορετική θέση στη λήψη αποφάσεων, στη διαχείριση των ε, project αντί να δώσουν τα χρήματα σε ένα οργανισμό των ΗΠΑ και εκεί και πέρα να τα ξεχάσουν. Γι' αυτό και τίθεται το ερωτηματικό το οποίο καμιά φορά βάζουμε εμείς. Δηλαδή ποιος είναι ο λόγος. Εμείς βρήκαμε ότι τα trust fund ανταποκρίνονται σε κατεπιδούς καταστάσεις. Το ερώτημα είναι λειτουργούν ως τέτοια. Συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά ως τέτοια και είναι δικαιολογημένα όπως με το Africa Trust Fund το οποίο άρχισε για κάποιο λόγο, μετά άρχισε να επεκτείνεται και μετά ε, άρχισε να επιλαμβάνεται τη μετανάστευση. Η μετανάστευση είναι καινούριο πρόβλημα. Ε, μέχρι πότε θα είναι καινούριο πρόβλημα. Και γιατί δεν αντιμετωπίζεται από την συνήθι χρηματοδότηση. Έχουν λοιπόν κάποια ερωτηματικά που ξεπηδούν σχετικά με τα Trust Fund. Και αυτό είναι και από τα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Και ποιο είναι και ο ρόλο συγκεκριμένα του Κοινοβουλίου. Εφόσον δημιουργούνται Trust Fund εκτό συνήθων διαδικασιών και εκτός συνήθων διαδικασιών και άλλων τμήματων του προϋπολογισμού. Εγώ είμαι ειδικευμένο στους προϋπολογισμούς, ιδίως στον εσωτερικό, αλλά έχω εξετάσει και κάποιους εξωτερικούς προϋπολογισμούς. Το ερώτημα εδώ είναι η διαχείριση, η governance. Μπορούν να μπουν μαζί αυτά τα πράγματα, η πίεση από τις έκτακτες καταστάσεις και να ενταχθούν μέσα στον μηχανισμό του προϋπολογισμού που έχουμε και στα κονδύλια που έχουμε διότι τα χρήματα περικόπτονται και μετά η λύση είναι να δημιουργηθούν εξωτερικά trust fund και κάποια στιγμή τα πράγματα που είναι συνήθι περιστατικά γίνονται πλέον emergencies γιατί δεν υπάρχουν πια αρκετά χρήματα και γίνεται μια εξωτερική κατάσταση και εκεί μπαίνεται πλέον στην δυσκολία, στο πρόβλημα. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι ορισμένα τμήματα του Africa Trust Fund δηλαδή υπάρχει αίσθηση ότι κάτι πρέπει να γίνει, ψάχνουν να βρουν κάποια χρήματα για κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν, όπως για παράδειγμα για τη μετανάστευση, η οποία έχει σχέση ίσως και με κάποια τοπική εξέλιξη που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Μετά χρησιμοποιούν διαδικασίε CDF και χρήματα από τον κανονικό προϋπολογισμό, αλλά έτσι εξεφεύγουν από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Και είναι και ένα ζήτημα ορθότητας. Δεν θέλω να δω τώρα μαζί σας όλες τις συστάσεις που έχουμε κάνει. Εμείς έχουμε εκφράσει μια ανησυχία σχετικά με το γεγονός ότι η ιδέα αυτή των καταπιστευμάτων, των Trust Fund, πάει να ξεφύγει λίγο από το χαρακτήρα της, της έκτακτης κατάστασης, της κατεπίγουσας κατάστασης και πάει να γίνει συνήθεια, πάει να γίνει ρουτίνα. Από τη στιγμή λοιπόν που περιορίζεται ο προπολογισμό, αυτή είναι η ανταπόκριση. Και το γεγονός ότι αυτό εμφανίζεται ως τάση και αλλού, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, όπου χώρες μέλη του προσπαθούν να ανακτήσουν κάπως τον έλεγχο των εξωτερικών δράσεων εκτός πλαισίων διεθνών οργανισμών. Και αυτό είναι ένα θέμα. Και ένα θέμα που είναι επίσης για μας σημαντικό είναι ποιες είναι οι αιτίες, ποιες είναι οι ρίζες αυτό επιτρέπει να ασκηθεί μια καλύτερη πολιτική, γιατί και το ζήτημα είναι βέβαια και η αποτελεσματικότητα. Είναι ταχύτερη έτσι η δράση, έχει περισσότερα αποτελέσματα. Για κάποια trust βλέπουμε πραγματικά λόγο να δημιουργηθούν. Το ζήτημα είναι βέβαια πώς συνεχίζεται η λειτουργία τους. Και το άλλο είναι, τέλος πάντων, πού βάζει κανείς το όριο και από πού θα πει από πού και πέρα θα πει όχι, δεν θα πρέπει να συνεχίσουν πάνω σε αυτή τη γραμμή, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε έτσι το ΑΒ θέμα βλέπουμε λίγο και το θέμα αυτό σαν μια προσπάθεια άσκησης εξωτερικής πολιτικής από κάποιες χώρες μέλη, το βλέπει αυτό κανείς και στη σχετική βιβλιογραφία, είναι μια πίεση, είναι ένα πρόβλημα που μπορεί ωστόσο να συμβεί και όταν πάει να κάνει κανείς εξωτερική πολιτική μέσω Trust Fund η ιδέα να υπάρχει ένας υπερεθνικός οργανισμός ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράδειγμα, ε, και δεν ταιριάζει μέσα σε αυτή την ιδέα Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα που έχουμε. Και βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εμείς προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε. Δεν προχωρούμε σε αξιολόγηση του πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά. Εξετάζουμε κάποιους θεμελιώδεις κανόνες ελέγχου και governance, διαχείρισης. Δηλαδή δεν αξιολογούμε, ούτε κρίνουμε τα ίδια τα trust fund. Εμείς εξετάζουμε μόνο αν οι διαδικασίες είναι σωστές και εμείς βρίσκουμε ότι σε κάποια σημεία θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Αυτά είναι λίγο πολύ τα θέματα. Να μην μπω σε όλα αυτά τα συμπεράσματα γιατί θα αναγκαστώ να μακρηγορήσω. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε και με άλλα trust fund. Τα ευρωπαϊκά ωστόσο είναι μοναδικά. Αλλά trust fund δεν έχουν όλα τον ίδιο χαρακτήρα ούτε έχουν δημοκρατικό έλεγχο από κοινοβούλιο. Βρήκαμε λοιπόν δύσκολο να τα συγκρίνουμε τα ευρωπαϊκά με άλλα trust fund και να μην συγχαίουμε τα trust fund με εκείνα τα οποία προβληθούν για παράδειγμα για την πολιτική γειτονία ή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πολλά από αυτά έχουν το ίδιο όνομα, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν τέσσερα emergency trust fund και άλλα με, άλλη, με άλλο χαρακτήρα. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δει κανεί ότι υπάρχει αυτό ο πολλαπλασιασμό των trust fund και εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάποια δυσκολία να κατανοήσει κανείς την λογική των trust fund και κυρίως να χρησιμοποιούν τα ίδια λόγια, τους, τις ίδιες λέξεις, τους τίτλους. Τους έχουμε το Africa Trust Fund και έχουμε και το Trust Fund for Africa. Το ένα είναι μηχανισμός δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το άλλο είναι Emergency Fund. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση να δω εάν έχουμε κάποια ιδιαίτερη σύσταση, με κάποια ιδιαίτερη σημασία δηλαδή. Ένα άλλο θέμα είναι, όπως λέχθηκε κιόλας, είδαμε σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες συμφωνίες, φαίνεται να υπάρχει μια προτίμηση για συνεργασία με κάποιες χώρες Και βλέπουμε επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διαφορετικά όργανα, Έχετε το governance body και το implementation body, αλλά σε αυτά η σύνθεση είναι ίδια, είναι τα ίδια πρόσωπα. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Όπου ανακατεύονται δηλαδή η δίψη αποφάσεων και η εκτέλεση, ή προτιμησιακές συνεργασίες με κάποιους κρατικούς οργανισμούς. Τους δίνεται η προτίμηση να συμμετάσχουν και μετά γίνεται ένα είδος συμπεγνία το οποίο ε, είναι πρόβλημα, δεν θα πρέπει να υπάρχει και έχουμε ανακαλύψει κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζουμε ότι υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου, δημοκρατικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάζω να δω μήπως έχω ξεχαστεί. Ποτέ τελευταίο, ίσως τελευταία σύσταση θα έλεγα είναι ότι βρήκαμε κάποια χρήσιμα στοιχεία, δηλαδή για παράδειγμα στα Ηνωμένα Έθνη έχουν πολλά trust fund και έχουν και αυτοί πρόβλημα με τα trust fund. Και εκεί δεν είναι απαραγμένοι προβλημάτων. Έχουν τουλάχιστον ένα πόρταλ, μία ε, πύλη και εκεί είναι πιο ενοποιημένα και έχουν ένα ενιαίο το οποίο ασχολείται με όλα αυτά τα trust fund εκεί μας φαίνεται σωστό γιατί δίνεται κάπως περισσότερη σαφήνεια και υπάρχει ένα single point of information, κάτι το οποίο διευκολύνει τα πράγματα και θα τα διευκόλυνε και αν εφαρμοζόταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θετικό παράδειγμα από τα Ηνωμένα Έθνη. Έρχονται βέβαια ορισμένοι και λένε ναι, αλλά κοιτάξτε και στα Ηνωμένα Έθνη δεν λειτουργούν τόσο καλά τα πράγματα. Ναι, αν όμως υπάρχει ένα καλό παράδειγμα, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς αυτό, δηλαδή να ανοίξετε κι εσείς μια ιστιακή πύλη και να, μια δικτυακή πύλη δηλαδή και να δείτε να δίνετε κι εσείς τις προφορίες αυτές και να έχουν και κάποιες εικονικές gateways για να μπορεί να μπαίνει κανείς να λαμβάνει τις προφορίες που θέλει τα οποία δεν βρίσκει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αρκεστώ σε αυτά. Εάν έχετε ερωτήσεις για το μέλλον των προϋπολογισμών κλπ. πολύ ευχαριστώ να προσπαθήσω να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη που σας έκανα να βιαστείτε, αλλά για να έχουμε λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις. Να σας πω, συνάδελφοι, ότι αύριο ε, έχει ε, ε, σύσκεψη το Συμβούλιο για το καταπίστημα της Αφρικής. Άλλαξαν την ημερομηνία, αλλά δυστυχώς είναι ταυτόχρονα με την Επιτροπή μας. Οπότε εγώ είμαι εδώ και ο Ινάτσιο Κοράο θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή μας στο καταπίστευμα αύριο. Βελτιωνόμαστε όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Και όταν κάναμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, είχαμε βουλευτές που συμμετείχαν στο ίδιο το καταστατικό. Στο παρελθόν, Συχνά ενημερωνόμασταν με κατόπιν εορτή. Και ήταν δύσκολο την πρώτη φορά, γιατί ήμασταν στις εκλογές το 2014 για το καταπίστευμα Μπέκου. Αλλά έκτοτε ε, ε, πάνε καλύτερα τα πράγματα. Συνάδελφοι, ξεκινάμε με την Τζούντι της Αργεντίνη, τον κύριο Σαφχάουζερ και την κυρία Χόιμπρουκ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το ΣΕΠΣ που έκανε αυτή την έρευνα. Η Επιτροπή μας επίσης στην εργασία της ιδιαίτερα Έχουμε μια νέα ομάδα εργασίας για τη μετανάστευση, ότι προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη για την αναπτυξιακή βοήθεια και τη μετανάστευση, να κατανοήσουμε καλύτερα τα σχετικά προβλήματα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε δει πιο, πιο μπροστά γιατί είναι επίγουσα η κατάσταση, έκτακτη ανάγκη και ρωτήσατε ποια είναι η έκτακτη ανάγκη. Όμως, εφόσον το καταπίστευμα έκτακτης ανάγκης εκπνέει το 2020, τότε τι θα γίνει. Γιατί τα project που έχουν ξεκινήσει συχνά ε, έχουν ξεκινήσει από μεγάλες, μεγάλους διεθνείς δωρητές ή ε, οργανισμούς αναπτυξιακής συνεργασίας που συνδέονται με ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Ενώ παλιότερα τα ίδια project μπορεί να γίνονταν με μικρούς τοπικούς ε, παράγοντες, φορείς της, της κοινωνίας των πολιτών στα αναπτυσσόμενες χώρες και έχω ακούσει τέτοιες διαμαρτυρίες ότι δεν συνεχίστηκε αυτή η χρηματοδότηση και ότι ε, δεν λέω, ας πούμε, για το GIZ, ε, το γερμανικό GIZ, ε, μπαίνει και παίρνει τη δουλειά. Ε, εμείς τι έχουμε κάνει με την ανάπτυξη της τοπικής υποδομής. Πώς συνδέεται αυτή όταν έχει τελειώσει το έργο ή όταν έχει τελειώσει ο χρόνος. Ο κύριος Σαφχάουζερ. Κύριε Σαφχάουζερ, ζητήσατε το λόγο. Ναι. Το έχω πει επανελειμμένα. Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ του Ταμείου. Όμως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας. Από την μια πλευρά έχουμε του ε, δημοσιονομική ε, ε, δημοσιονομικά κονδύλια τα οποία καταλήγουν κάπου στη μαύρη τρύπα του κρατικού προϋπολογισμού. Και μετά έχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια που πάει προς τις ΜΚΟ. Χρησιμεύει γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ σε έκτακτε καταστάσεις. Πρέπει να βοηθηθούν οι πληθυσμοί ακόμα και όταν δεν υπάρχει πια κράτος. Δεν είναι αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά πρέπει να κάνουμε ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Μετά υπάρχει αναπτυξιακή βοήθεια ε, βοήθεια και για την ασφάλεια. Αυτό δικαιολογεί τις νέες πολιτικές. Είμαστε ενώπιον νέων καταστάσεων όπου η ασφάλεια συνδέεται με την ανάπτυξη. Γι' αυτό χρειάζεται ένα κατάλληλο μέσο. Το μέσο του καταπιστεύοντος είναι καλό με την προϋπόθεση ότι συνδέει τα δύο θέματα ασφάλεια και ανάπτυξη και τα προσεγγίζει από εκείνου Δεύτερον, ότι θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με το εκάστοτε κράτο, να υπάρχει μια συναπόφαση. Οι δυο πρέπει να υπογράφουν. Από τη μια πλευρά το κράτο και από την άλλη εκπρόσωπο τη Ένωση επιτόπου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν πάμε σε έναν γενικό προπολογισμό, πάμε άμεσα προ projects ασφάλεια κάθετο ανάπτυξη που θα πρέπει να εξασφαλίζουν δηλαδή την ασφάλεια και θα δημιουργούν ε, δυναμικές οικονομικές ανάπτυξης. Και αυτό το μέσο, το καταπίστευμα Μπέκου και το τωρινό καταπίστευμα δεν το επιτρέπουν γιατί δεν γίνονται σε συνεργασία με το κράτος. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει βεβαίως το Κοινοβούλιο να μην είναι εκτός όλων αυτών. Δεν πρέπει να κάνουμε εκ έξτρα προπολογισμό, γιατί έτσι παρακάμπτεται το Κοινοβούλιο, παρακάμπτονται οι διαδικασίες χρηματοδότησης της Κομισιόν και εννοείται ότι το σύνολο της οικονομικής διαχείρισης πρέπει να είναι υπό ε, ε, διαχείριση ή υποεποπτεία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάνουμε μια επενδυτική προσπάθεια ότι γινόμαστε ανεύθυνοι. Όχι. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέσο. Δηλαδή ανάπτυξη και ασφάλεια με τα αφρικανικά κράτη. Αλλά όχι να πηγαίνει στη μαύρη τρύπα τα χρήματα αυτά του δεκάστοτε εθνικού προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Χόιμπρουκ. Σας ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς τους δυο για την εκθεσή που δεν πρόλαβα να την παρακολουθήσω όλοι. Τα όσα άκουσα όμως ε, βρίσκω ότι ανταποκρίνονται απολύτω και στην κριτική που ασκούμε εμείς συχνά. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα χρήματα ε, δεν υπόκεινται πάντοτε στον ελεγκτικό μας ρόλο. Είπατε και εσείς ότι καμιά φορά καταστρατηγείται η αρμοδιότητα αυτή του Κοινοβουλίου και ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν φαίνεται να είναι εντάξει. Από τη δική μας πλευρά έχουμε ασκήσει κατ' επανάληψη κριτική του είδους αυτού την χρηματοδότηση. Η ερώτησή μου είναι τώρα, έχετε εξετάσει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα αυτά στο μέλλον και ιδίως ό,τι αφορά τους ενιαίους μηχανισμούς, single instrument, το οποίο ε, θα ήθελε να εντάξει στον μελλοντικό χρηματοδοτικό σχεδιασμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μένα φαίνεται να διαγράφεται κάπως, ε, εφόσον έχουμε ένα τέτοιο εξωτερικό μηχανισμό με 20% ευελιξία, ότι μέσα σε αυτό το 20% ευελιξία, flexibility, μπορούν να μπουν πάρα πολλά πράγματα. Και αυτά που παίρνουν τώρα μέσα από trust fund και τα οποία υποτίθεται ότι είναι χρονικά περιορισμένα. Έχετε εξετάσει λοιπόν το θέμα προς την κατεύθυνση αυτή του μέλλοντος ή έχετε δει μονά, μονάχα το πώς λειτουργούν έως τώρα με, το, με τον τρόπο που είναι οργανωμένα αυτά τα trust fund έως τώρα. Αυτό σημαίνει και το τέλος τώρα των ερωτήσεων. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Ένας λόγος που επικαλείται συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Trust Fund είναι ότι λέει ότι μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι. Έχετε κάποια εκτίμηση πόσο έχουν συμβάλει άλλοι χώρες μέλη, άλλες τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμοί και σας δίνω και πάλι το μικρόφωνο. Okay, I will, I will. No, we'll let them respond, then we'll let the ναι, θα τους δώσουμε το λόγο να απαντήσουν και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Προϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Μιλάω πολλές γλώσσες, αλλά θα σας απαντήσω στα αγγλικά. Λοιπόν, για τις ε, προοπτικές από εδώ και πέρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι είναι αποκλειστικό ζήτημα της αναπτυξιακής βοήθειας. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα μέτρο ε, έκτακτης ανάγκης, ε, αναπόφευκτα είτε διονύζεται είτε εξαφανίζεται. Κλείπει και όλοι ξαφνικά διαμαρτύρονται. Είναι σημαντικό κάποιος το σημαντικό δυνατόν να αρχίσει να αναλύει και να ε, βλέπει πώς μπορεί αυτό να επιστρέψει στην κοινωνία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι όταν πρέπει να δράσει κανείς πολύ γρήγορα σε ένα project, ε, να θέλει ε, να απευθυνθεί στους συνήθεις εταίρους, αν αυτό είναι κατάλληλο δός, σε ορισμένες περιπτώσεις. Μετά όμως θα πρέπει να υπάρχει μια μεθοδολογία αυτό θα πρέπει ε, να το δει κάποιος και δεν το βλέπω συχνά από την αρχή. Δηλαδή εντάξει, έστω ότι θεσπίζεται ένα ε, τέτοιο ταμείο καταπηγόντως, αλλά πρέπει να δούμε μετά τι, πώς θα συνεχιστεί αυτή ε, η δραστηριότητα και ποιος θα την αναλάβει. Αυτό είναι σοβαρό κατά τη γνώμη μου. Ρωτήσατε επίσης ε, ποια είναι η χρησιμότητα του Ταμείου. Σαφώς και εμείς δεν θέτουμε τέτοια ζητήματα όταν υπάρχουν θέματα ασφάλειας, ανθρωπιστικών κρίσεων. Μπορεί να υπάρχει ένα καταπίστευμα όταν δεν υπάρχει άλλη ευελιξία. Και αυτό είναι άλλο ερώτημα. Γιατί ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό δεν έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί χωρί ε, να χρειάζεται να θεσπιστεί εξωτερικό ταμείο. Αν γινόταν αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο ε, για τέτοια ζητήματα, ιδίω για την ασφάλεια. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη με ζητήματα που προηγουμένως με, που, με την συνήθεια αναπτυξιακή βοήθεια δεν υπήρχαν. Είναι πιο περίπλογη η κατάσταση πλέον. όπως και ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν ε, σχεδιασμένος για περιπτώσεις κρίσης, όπως είδαμε, ούτε και εξωτερικά όμως. Δεν ήταν ε, σχεδιασμένο σωστά για να αντιμετωπίζει κρίσει. Το θέμα είναι κατά πόσο τώρα μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν προπολογισμό που θα έχει αυτή τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε κρίσει χωρί να μπαίνει σε όλε αυτές τι δεδαλώδες διαδικασίε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πρώτον, υπήρχε το θέμα για τις χώρες που συμμετέχουν. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά για, για άλλα θέματα ε, αναπτυξικής βοήθειας υπάρχουν ε, δομές διακυβέρνησης, ακόμα και στο λεγόμενο blending, και τα καταπιστεύματα με την ε, Τράπεζα Επενδύσεων και όπου εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνήθως οι χώρες ε, συμμετέχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό. Θα μπορούσε λοιπόν να ακολουθηθεί το ίδιο παράδειγμα και εδώ. με μάλιστα μπορώ να σας πω που βλέπω τέτοια στοιχεία. Τώρα για τον ενιαίο μηχανισμό. Υπάρχει γενικά μια τέτοια τάση θέσπισης ενιαίων μηχανισμών και αυτό μπορεί να προκύπτει ως απόρριτο γεγονότος ότι έχουμε υπερβολικό αριθμό μέσων. Από την άλλη, είναι ένας τρόπος ε, να κινητοποιήσουμε πιο γρήγορα τη χρηματοδότηση, γιατί δεν ε, απαιτείται αδειοδότηση μας δίνει λοιπόν αυτό ευελιξία, μπορεί να δημιουργήσει όμως και προβλήματα γιατί δεν μπορεί κανείς ε, να ε, εγγυηθεί την ε, σταθερότητα αυτών των τομέων αλλά το ποσοστό του 20% ευελιξίας θα μπορούσε να λύσει κάποια ζητήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο φτάνει η ευελιξία ή αν πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό που δεν θα κατανέμεται προηγουμένως. Γιατί υπάρχει διαδικασία αφαίρεση κονδυλίων από ένα μέσο και διοχέτευση σε έναν άλλο. Είδαμε λοιπόν ότι κόβουμε χρήματα από την έρευνα και ανάπτυξη για, για να μην έχουμε περικόπες στη γεωργία. Αυτό που έχω ζητήσει και εγώ και άλλοι είναι να υπάρχει κάτι το οποίο να χρηματοδοτείται σταθερά και ε, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί εάν υπάρξει μια τέτοια ανάγκη. Μετά, η συνεισφορά των χωρών. Γενικά, τα καταπιστεύματα δεν προσελκύουν ε, χρηματοδότηση πολλών κρατών μελών. Συνήθως πρόκειται έτσι για συμβολικά ποσά, απλά και μόνο για να μπει το όνομα της χώρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην πορεία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, επαναδιοχετεύσει χρήματα από το ενωσιακό προπολογισμό για να καλύψει ζητήματα που δεν θα τα κάλυπταν κράτη-μέλη. Και αυτό υπάρχει σχεδόν σε όλα τα καταπιστεύματα. Από τις ε, προσδοκίες ε, του σχεδίου Juncker, ότι ότι θα υπάρχει αυτός ο μηχανισμός ε, και με χρηματοδότηση των κρατών μελών, αλλά γενικά βλέπουμε ότι δεν είναι σημαντική η συμβολή των κρατών μελών, εκτός και αν πρόκειται για την χώρα που ξεκίνησε την όλη πρωτοβουλία. Όμως και πάλι η χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής. Γενικά δεν είναι εξαιρετική η συνεισφορά των κρατομελών στη χρηματοδότηση των καταπιστευμάτων. Ναι, να σα δώσω κι εγώ μερικά στοιχεία. Για το καταπίστευμα Μπέκου, τα τρία τέταρτα τη συνολική χρηματοδότηση προέκυψαν από τον ενωσιακό προπολογισμό και μόλι το ένα τέταρτο από τα κρατημέλη. η χρηματοδότηση των κρατών μελών ήταν ακόμα μικρότερη σε σχέση με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε, ό,τι αφορά το καταπίστευμα για την Αφρική. 3,38 δις είχαν δεσμευτεί συνολικά, 2,9 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλις 400 εκατομμύρια από τα κράτη-μέλη και άλλους δωρητές. Υπάρχει λοιπόν προσθετικότητα και τα κράτη-μέλη λαμβάνουν αυτή την προβολή, όμως, όπως είπε και ο Χόρχε, υπάρχει δέσμευση από τα κράτη-μέλη, υπάρχει και προσδοκία από τα κράτη-μέλη να το υλοποιήσουν. Και από μία διαδικτυακή έρευνα που κάναμε και από συζητήσεις σε focus group, είδαμε ότι οι οργανώσεις εκφράζουν ξεκάθαρα ε, αυτή τους ε, τη δυσαρέσκεια. Κάτι άλλο είναι ότι υπάρχει αυτό ο κανόνα του 5% ότι μόλις το 5% των καταπιστευμάτων μπορούν να διοχετευθούν. Γι' αυτό προέκυψε και όλο το συμπέρασμα ότι τα ενωσιακά καταπιστεύματα θα είναι φτηνότερα, πιο οικονομικά από, τα, από αυτά του ΟΗΕ. Όμως και στη διαχείρισή τους βλέπουμε τι δεν συμπεριλαμβάνεται στα διοικητικά κόστη. Αυτό το θέμα το έθιξε και το ελεγκτικό συνέδριο. Και από όλη τη διαδικασία είδαμε ότι αρκετά συχνά ε, λαμβάνουν τα κονδύλια εναπτυξιακέ ε, υπηρεσίε ε, των κρατών μελών, αλλά δεν είναι επιχειρησιακό το έργο, οπότε αναθέτει σε κάποιον άλλον οργανισμό και τότε ο άλλος οργανισμός το αναθέτει εξωτερικά σε κάποιο στο επίπεδο. Τι λοιπόν ζήτημα εποπτείας, διαχείρισης, αλλά και το ζήτημα κατά πόσο ο τρόπος που υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα είναι ο πιο οικονομικά αποδοτικός. Από τον Μπεκού βλέπουμε ότι όπου υπάρχει περιορισμός ε, στον ανταγωνισμό, τα προγράμματα πιο γρήγορα ε, διοργανώνονταν και υλοποιούντο. Υπήρχαν πιο αξιοκρατικά κριτήρια, ας πούμε. Ζητώ συγγνώμη, λέει πρόεδρος, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Um, um yeah, please, Commission, European Commission, is Παρακαλώ, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, συνοπτικά σε όλες τις παρατηρήσεις και προτάσεις και συστάσεις. Καταρχά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη μελέτη και για την προστιθέμενη αξία της μελέτης. Είναι πάντοτε πολύ σημαντικό να βλέπουμε όλα αυτά ε, για την Κομισιόν. Για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζουμε τη συμμετοχή ε, του Ευρωκοινοβουλίου στη διαχείριση αυτών των ταμείων. Ε, το Κοινοβούλιο έχει θέση εποπτική στο Διοικητικό Συμβούλιο του Καταπιστέματος για την Αφρική και μάλιστα καθορίζει και έτσι η επόμενη συνεδρίαση, το είπατε και εσείς ίδια πρόεδρε, για να μπορεί να συμμετέχει εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου είναι σημαντικό για τη δράση να αναφέρουμε ότι η υλοποίηση του προπολογισμού είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο δημοσιονομικό κανονισμό προβλέπει μάλιστα ότι τα καταπιστεύματα είναι μέσα εφαρμογή και υλοποίηση του προπολογισμού στον τομέα τη εξωτερική δράση. Γι' αυτό το λόγο η διαδικασία λήψη απόφαση για την υλοποίηση των καταπιστευμάτων παραμένει αρμοδιότητα τη Κομισιόν, όμω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εφαρμόσει το δικαίωμα ε, παρακολούθησης μέσω μιας μηνιαίας έκθεσης για την υλοποίηση κάθε ταμείου Κάθε καταπιστεύματος είναι ένα έγγραφο το οποίο ε, συντάσσει η δεζε, Budge, η Γενική Διεύθυνση για τον Προϋπολογισμό και τριμηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες κάθε καταπιστεύματος. Τώρα μιλήσαμε για την ευελιξία και την προστιθέμενη αξία των ε, ε, καταπιστευμάτων. Το καταπίστευμα για την Αφρική θέλει να δώσει γρήγορες και ευέλικτες απαντήσεις, αλλά και αποτελεσματικές απαντήσεις σε εκτακτές καταστάσεις. Ε, αστάθεια στο Σαχέλ και το Τσάντο, που είναι πήγου η κατάσταση, και ε, μεταναστευτική κρίση. Είναι αλήθεια ότι η μελέτη δεν αφορούσε ε, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, αλλά να θυμίσω πως αυτό το καταπίστημα επέτρεψε να σωθούν 3.700 άνθρωποι στο ενέρημο του Νίγηρα και ακόμη τόσοι υποφελήθηκαν από τις υπηρεσίες επιστροφής της χώρας περιληψής τους. Αυτά είναι τα επιτεύγματα. Με την κλασική ε, αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε καταφέρει αυτό. Πρέπει να είναι αυτό ε, μεταξύ μας σαφές. Αναγκαστικές ε, τώρα, αναγκαστικοί εκτοπισμοί Υπάρχουν, ναι, η αποστολή στην ε, Σενεγάλη έδειξε πως υπάρχουν project που λειτουργούν και είναι αλήθεια πως έχουμε χρησιμοποιήσει αποδοτικά προγράμματα που υπήρχαν ήδη και λειτουργούσαν στα κράτη-μέλη, από, δηλαδή από οργανισμού των κρατών μελών με στόχο την ευελιξία και την αποδοτικότητα. Το Κοινοβούλιο επισκέφθηκε αυτά τα project και ήδη έχουμε αποτελέσματα. Αν έπρεπε να κάνουμε μελέτες εντοπισμού τη διατύπωση του προγραμμάτων για τα project αυτά, δεν θα είχαμε ήδη αυτά τα αποτελέσματα, όπω αυτά που είδατε στη Σενεγάλη. Αν αναλύσει κανείς σύντομα τις προθεσμίες ανάμεσα στο καταπίστευμα για την Αφρική και τα, τα, αποτελέσματα των ταμείων της, ε, του ΦΕΔ και της ε, Ένωσης, ε, θα δούμε ότι η λειτουργία του καταπιστεύματος είναι πολύ πιο γρήγορη. 33 μέρες κατά μέσο όρο, ενώ 300 για τα άλλα μέσα και 180 για τις συμβάσεις. Χρειάζονται 174 μέρες μεταξύ για τα μέσα του ΦΕΔ και του προϋπολογισμού, δηλαδή του Ταμείου για την Ανάπτυξη. Ε, είναι πολύ πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Τώρα, ο ρόλος των κρατών μελών για ενημέρωσή σας υπάρχει έλεγχος ελεκτικού συνεδρίου που τρέχει και που δεν έχει δείξει σύγκρουση ε, συμφερόντων από πλευρά των κρατών μερών. Αυτό μέσα στο πλαίσιο του συμβασμού του δημοσιονομικού κανονισμού. Μόνο οι εκπρόσωποι των κρατών μελών έχουν δικαίωμα ψήφου και αυτό στο, είναι μέσα στο πλαίσιο του, συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμένοι από αυτούς τους φορείς συμμετέχουν ως παρατηρητές μόνο της Κομισιόν. Είναι αλήθεια πως ορισμένοι οργανισμοί λαμβάνουν ε, σημαντικά χρήματα, σημαντικά ποσά. Γιατί, Γιατί είναι παρόντες τόπου περισσότερο από άλλους, έχουν σημαντικά μέσα να εφερμόσουν και έχουν μια πραγματική προστιθέμενη αξία σε σχέση με το καταπίστευμα και άλλοι φορεί πρέπει να λειτουργήσουν επιτόπου. Ενώ ένα οργανισμό ή μια ΚΕΟ να πάει εκεί επιτόπου πρέπει να βρει γραφεία, να καταλάβει τη χώρα. Όλα αυτά παίρνουν χρόνο. Εδώ βρισκόμαστε σε έκτακτε καταστάσει που δεν θέλουμε να πούμε γρήγορα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα οργανισμό να, φτιάξει, να πάρει δύο-τρία χρόνια ώστε να στηθεί σωστά επιτόπου. Αντίθετα, ε, αυτό δεν σημαίνει πω καταργούνται αυτοί οι οργανισμοί. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε μαζί τους αλλά ε, όταν θέλουμε γρήγορα να, κάνουμε, να συνάψουμε συμβάσεις και να ε, υλοποιήσουμε τα project δεν ήταν δυνατόν να περιμένουμε μήνες και χρόνια μέχρι ότου στηθεί κάποιο ε, οργανισμός ε, και να πάρει την εικόνα της κατάστασης. Οι έξι συμβάσεις στις 10 εφαρμόζονται, υλοποιούνται από οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών. Όταν μιλάμε δηλαδή για κοινωνία των πολιτών, σημαίνει για σημαντικό κομμάτι του καταπιστέματος μέσω των κονδυλίων που πάνε άμεσα στην κοινωνία των πολιτών και μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των υπηρεσιών των κρατών μελών μας, πάνω από το ίμιση του καταπιστέματος εφαρμόζεται από τη Διεθνή Κοινωνία των Πολιτών και την τοπική κοινωνία των πολιτών. Για να επανέλθουμε τώρα σε σχέση με τα κράτη που συμμετείχαν με 400 ε, εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να δούμε μισογεμάτο μισάδιο το ποτήρι. Είναι αλήθεια ότι η Κομισιόν θα ήθελε να προσθέσουν τα κράτη μέλη άλλα 4 δι. Το έχουμε πει ξανά και ξανά. δυστυχώ αυτό δεν έχει ακόμα συμβεί. Πιστεύουμε ότι πως ήδη τα 400 εκατομμύρια είναι μια σοβαρή προσπάθεια. Ειδικά αν δούμε και εδώ έχω τα τελευταία στοιχεία που θα παρουσιαστούν αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γερμανία είναι στα 157 εκατομμύρια, η Ιταλία στα 104, αλλά η Τσεχία ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια, η Δανία 10, η Πολωνία 10, οι κατοχώρε 26, η Γαλλία 9 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ ε, κάτι έχει αντιστραφεί. Υπάρχουν χώρες ε, όπως η Πολωνία που Ε, ξεπερνούν τη Γαλλία <laughs> αυτό το καταπίστευμα. Κάτι έχει αλλάξει. Να αναφέρω ε, επίση το ε, ΝΟΙΕ και το καταπίστευμα του ΟΗΕ. Τι, έχουν επιτρέψει αυτά τα καταπιστεύματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην βάζει τα χρήματά της σε καταπιστεύματα του ΟΗΕ, όπου εκεί δεν θα συζητούσαμε αν το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να έχει τον έλεγχο δικαίωμα ελέγχου. Όλα αυτά γίνονταν παλιότερα, όχι πλέον. Γιατί χάρη στα καταπιστέματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται αυτή η συζήτηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω ως Ευρωπαίος πολίτης, το Ευρωκοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει, να επιβλέπει. Αυτό είναι δυνατόν λόγω των ευρωπαϊκών καταπιστευμάτων, της ύπαρξης αυτών. Και να προσθέσω κάτι ακόμα. Τα καταπιστεύματα έχουν μία συνοχή δική τους. Θα ήταν ζημιογόνο να δημιουργηθεί μία παράλληλη δομή με μόνο καταπιστεύματα που δεν θα εντάσσονται στο πολιτικό διάλογο και τις ε, ε, γεωγραφικές στηρίξεις ε, ρίσματα των κλασικών μέσων. Η συνοχή ανάμεσα στα κλασικά αναπτυξιακά μέσα και τα καταπιστεύματα είναι ουσιώδου σημασία. Στην DG ή DG όλα αυτά τα καταπιστέματα είναι σημαντικό να, ε, ε, να είναι ε, ολοκληρωμένα με τις αντιπροσωπείες μας αλλά και με τις γεωγραφικές μονάδες ή τμήματα. Και άλλες ερωτήσεις. Κύριε Σαφχάουζερ, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πω θέλω μόνο ότι... Sorry, with the whole... Sorry, so who's speaking on the phone, please? Please, we can all hear you. Συγγνώμη, μη μιλάτε στο τηλέφωνο γιατί σας ακούμε όλοι. <laughs> Λοιπόν, τα, χρήμα, τα κράτη συμβάλλουν διμερώς χρήματα. Πώς ξέρουμε πως αυτό δεν βγαίνει από τη διμερή τους βοήθεια και αν πρέπει να τα δαπανίσουν σε project και Πώ ελέγχονται. Και υπάρχουν ένα σωρό ερωτήματα. Και γιατί παίρνει τόσο χρόνο για να μπουν αυτά τα χρήματα στα κανονικά προγράμματα. Αυτά όλα πρέπει να συζητηθούν και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. Σα ευχαριστώ όλους, την Κομισιόν, τους προσκεκλημένους μα και σημαίνει βεβαία ότι θα επανέλθουμε συντόμω. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Εγώ ήξερα για έναν εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Ε, από πού είστε εσείς? Ναι. near? Όχι, ε, να αφήσουμε τότε τους διερμηνείς να φύγουν, λέει η Πρόεδρος. Είναι πολύ αργά, πρέπει να, πρέπει να κλείσουμε. Ε, λυπούμε, ελάτε εδώ να μου πείτε τι θέλετε, γιατί οι συνάδελφοι πρέπει να φύγουν. Αύριο στις 9 με τους συντονιστές και ψηφίζουμε στις 10 και 4.